Καλημέρα. Η Επιτροπή σήμερα θα καταφέρει να συνθέσει, να συγκροτήσει Προεδρείο. Οπότε θα βγούμε από αυτή την πολύ διόμορφη κατάσταση που ήμασταν μέχρι τώρα. Και βέβαια στο Προεδρείο προβλέπεται πρέπει κανονικά να υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες. Πριν περάσουμε λοιπόν στην εκλογή των αντιπροέδρων, να επιβεβαιώσω την ταυτότητα των αναπληρωματικών μελών. Θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να μας ε, γνωστοποιήσουν τα ονόματα των ε, αναπληρωτών. Σήμερα λοιπόν το πρωί έχουμε τον Γιώ Λάινεν που αντικαθεί την κυρία Χόφμαν, τον Καμπρίλε Πρέσ που αντικαστά την κυρία Μούντι, τον 50 Θηλβάγκα που εξ... αντικαστεί κυρία Μυριάντα και η κυρία Χάουταλα αντικαθιστά την κυρία Βά. Έχουμε λοιπόν τους αναπληρωτές που σας προνέφερα, με τους οποίους πιστεύω ότι έχουμε και απαρτία, <coughs> δηλαδή λάχιστο αριθμό 11, βουλευτές είναι παρόντες. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή των μελών του Προεδρείου από τον Ιανουάριο. Το Προεδρείο συγκριτά από τον Πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κ. Σαρβάμα. Οι πολιτικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία. Au terme duquel με βάση την οποία υποψήφιο για τη θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου κύριο Γκάιερ, για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου κύριο Μούρεσαν και για τη θέση του τέταρτου η κυρία Χολ Μάιερ. Κύριε Γκάιερ, είστε πραγματικά υποψήφιο. Είναι υποψήφιο. Το επιβεβαιώνει ο κύριο Μούρεσαν και αυτό. Κυρία Χολ Μάιερ, επίσης. Να ψηφίσουμε με μυστική ψηφοφορία ή νομίζω ότι μπορούμε να εκλέξουμε διαβόηση τους ε, τρεις υποψηφίους. Διαβοής λοιπόν. Je déclare donc. Επομένως, ε, ο Γιάννης Γκάιερ εκλέγεται στη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Στη θέση του τρίτου αντιπροέδρου ο Ζίγκρβιτ Μούρεσαν και στη θέση της τέταρτης αντιπροέδρου η Μόνικα Χολμάιερ. Καλό την κυρία και τους κυρίους αντιπροέδρους να έλθουν να καθίσουν στο Προεδρείο. Επίσης, έχω να σας προτείνω μία τροποποίηση σε μια διάταξη η οποία προβλέπει τη συζήτηση των εγγύσεων για τις εξωτερικές δράσεις ως πρώτο σημείο, αλλά για προσωπικούς λόγους, κύριε Χολμάιρ θα ήθελε τώρα να περάσουμε στη δική της έκθεση για την κτηριακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως για το Frontex, τη μέτρα του Frontex. Ähm, ähm, Κύριε Πρόεδρε, αποφασίζαμε την ε, Δευτέρα γιατί υπάρχει νομοδότηση για το θέμα αυτό σε σχέση με την ε, περαιτέρω ενοικίαση του κτίριου που θέλουμε να επιμηκυνθεί για να καλύψουμε αυτή την ε, επιμήκυνση χρειάζεται οικονομική ενίσχυση και θα πρέπει να το δούμε το συντομότερο δυνατό, γιατί μιλάμε για δύο κτίρια, για τον ίδιο σκοπό και για το ίδιο προσωπικό. Δύο χρόνια ενίκιο παραπάνω είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό. wir am Montag entscheiden würden για να το αποφασίσουμε τη Δευτέρα παραλαμβάνω. Θα ήθελε κάποιο το λόγο. Personne. Merci, Madame la... Ουδής, ευχαριστώ την κυρία Αντιπρόεδρο, την οποία και συγχαίρω εκ νέου. Και Ζητώ τώρα από την Ίντερ Γκαρθιά Θάμπαλ να μας παρουσιάσει την δική της έκθεση για το Ταμείο Εγγύσεων για τις εξωτερικές δράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγομαι. Θα μιλήσουμε λοιπόν ε, για την ΕΤΕ, για την, εξωτερική εντολή, την εντολή για τις εξωτερικές δράσεις Ήδη έχουμε ακούσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία παρουσίασε σε μια πρώτη φάση ποιε ήταν οι τροπολογίε, τροπολογίε που έχω καταθέσει και εγώ ω εισηγήτρια και θα ήθελα λοιπόν να αξιολογήσω και τι υπόλοιπε τι οποίε έλαβα και να δούμε σε ποιε μπορούμε να βρούμε κάποια συμφωνία. Τη στιγμή που, θα, που παρουσιάσαμε, συγχωρείτε, την ε, έκθεση, συνόψισα την γραμμή που ακολουθούμε σε πέντε κομμάτια. Πρώτο είναι το τμήμα με τα νούμερα, όπου υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία στο να αυξήσουμε την, ε, την κορυφή της πιθανής ε, ε, του πιθανού προπολογισμού, αλλά εδώ έχουμε κάποιες βασικές διαφορές μεταξύ σοσιαλιστών και ΕΛΚ, έτσι ώστε όλα αυτά τα πλαφών να συμφωνηθούν με έναν τρόπο που θα μας ικανοποιεί όλους. Να τροποποιήσουμε λοιπόν τους προϋπολογισμούς που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν για να αυξήσουμε τα κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα και για να μεταρρυθμίσουμε τους χώρους τους οποίους η ΕΤΕ έχει εκτελέσει ήδη τα έργα και έχει προ, ε, προκαταβάλει τα, τις δαπάνες, κυρίως δηλαδή στις χώρες μας που, της ανατολικής γειτονίας. Να σας πω λοιπόν πως εκεί καταλήξαμε σε μια έλλειψη ισορροπίας, ε, με μια μη ε, ισόρροπη συμμετοχή τις έτες στην Ανατολική Ευρώπη, ε, χαμηλότερη από ό,τι στην Νότια Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Ακόμα και αν διατηρήσουμε λοιπόν ε, το μεγαλύτερο κομμάτι ε, αυτών των κονδυλίων που διατίθονται για τις ανατολικούς μας γειτονές θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι για την ε, Νότια Ευρώπη και να προσθέσουμε και κάτι λιγότερο για την Λατινική Αμερική γιατί έχουμε μεταναστευτικές ε, πιέσεις όχι μόνο από τα ανατολικά μας σύνορα αλλά και από τα νότια και νομίζω ότι αν τροποποιήσουμε τα, το κανονισμό εδώ για την ΕΤΕ θα βοηθήσουμε χώρες που υπάρχει περισσότερη μετανάστευση και θα λάβουμε υπόψη και τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, για να τα χαρακτηρίσω έτσι, δηλαδή τι σημαίνει η νίκη Τραμπ στη ΣΥΠΑ και τι συμβαίνει όταν κλείνουν τα σύνορα εκεί, όπως επίσης το ότι έχει εγκαταλειφθεί η Λατινική Αμερική στην ε, ε, εξίσωση αυτή. Θα ήταν καλό λοιπόν να συνεχίσουμε να ε, εξετάζουμε τι γίνεται πέραν της δικής μας γειτονιάς. Ξέρω ότι είναι πιο κοντά σε εμάς αλλά νομίζω ότι όταν συμβαίνει και σε άλλες περιοχές του κόσμου πραγματικά ε, επηρεάζει την κατάσταση. Να επιστρέψουμε λοιπόν στην Λατινική Αμερική γιατί κάπου την έχουμε ξεχάσει. Σε, γενικούς, ε, σε γενικές γραμμές ε, συμφωνούμε. Θα διατηρηθεί αυτή η αύξηση που έχει στην πρόταση της Κομισιόν, αλλά νομίζω στην κατανομή θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή προσπάθεια για να καταλήξουμε σε κοινή θέση εδώ στην Επιτροπή μας. Το δεύτερο μπλοκ τροπολογιών που παρουσίασα έχουν να κάνουν με το νέο στόχο 4. Εγώ θέλησα να αλλάξω εδώ τη διατύπωση και να μην μιλάμε μόνο για μάχη κατά των ουσιαστικών λόγων που δημιουργούν την μετανάστευση, την, ε, τις αιτίες δηλαδή, γιατί λογικό είναι να ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε για ε, μάχη κατά των ε, γεννησιουργών αιτιών, αλλά να διευρύνουμε κάπως τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε και να βοηθήσουμε και τις χώρες αυτές να αναπτυχθούν και έτσι ο πληθυσμός του στη χώρα αυτή να μπορεί να ζει κανονικά και να μην αισθάνεται την ανάγκη να ξεκινήσει ένα ταξίδι ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο αντικατοπτρίζω αλλάζοντα το στόχο αυτό είναι και να δω πώς θα σας το εξηγήσω. Ότι η μετανάστευση αποτελεί συνέπεια των όσων συμβαίνουν στις χώρες αυτές και ότι είναι πολύ πιο λογικό αντί να αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις, να ε, αντιμετωπίζουμε τα αίτια. Και νομίζω είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση των όσων συμβαίνουν στις χώρες αυτές. Και αυτή η αντιμετώπιση είναι πιο σωστή από το να πάμε απλώς να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες, δηλαδή τη μετανάστευση. Επαναλαμβάνω, πως όταν επενδύουμε στις χώρες αυτές και βοηθάμε τις χώρες αυτές να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο, ο στόχος ο οποίος βρίσκεται πίσω από όλες αυτές τις πολιτικές και εδώ και στην εξωτερική ε, εντολή της ΕΤΕ, αλλά νομίζω ότι και αργότερα, γύρω στις 5.30, θα μιλήσουμε για την βιώσιμη ανάπτυξη και το σχετικό Ευρωπαϊκό Ταμείο, το οποίο ε, ουσιαστικά στους ίδιους στόχους ε, σκοπεύει. Είναι δηλαδή ε, μια βοήθεια προς αυτές για να αναπτυχθούν έτσι ώστε να προσφέρουν κάποιο είδους ε, μέλλον και ιδίω στον πιο νέο τους πληθυσμό που αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία δυνατότητα απασχόλησης. Αυτές είναι οι τροπολογίες και νομίζω με λίγο ε, καλή θέληση και δεξιοτεχνία θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ πολιτικών ομάδων και δεν θα πρέπει εμείς να εστιάζουμε μόνο στη μάχη κατά των συνεπειών αυτών των προβλημάτων που είναι η μετανάστευση, αλλά να το δούμε πιο γενικά. Το τρίτο μπλοκ τροπολογιών έχει να κάνει με τις πολιτικές για το φύλλο. Και πρέπει να σας πω πως χάρηκα που καταθέσατε τόσες πολλές τροπολογίες σχετικές έτσι ώστε να ελέγχουμε τις συνέπειες σε επίπεδο ισότητας μεταξύ ανδρών και γενιών. Πολλές ομάδες πολιτικές κατέθεσαν τέτοιου είδους τροπολογίες. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να συμφωνήσουμε τη διατύπωση και τη φρασιολογία. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να προσέχουμε να μην καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί όπου έχουμε να λάβει δράση. Πολλές τροπολογίες σχετικέ έλαβα και επαναλαμβάνω, συμφωνώ. Συμφωνώ απλώ να καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο. Και έχουμε και το άλλο μπλοκ τροπολογιών που έχει να κάνει με φορολογικός παραδείσους, φόρο απαλλαγή, φόρο διαφυγή, ε, φόρο αποφυγή, με συγχωρείτε. Και νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά και εδώ πάλι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είναι μια κοινή συμφωνία για το πώς θα το πούμε. Ένα τελευταίο θέμα στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το επόμενο, αλλά τα συζητάμε μαζί. Είναι μια θα έλεγα μεγάλη πλειοψηφία, δεν μπορώ ενδεχομένως να μιλήσω για συνένεση, στην Επιτροπή μας, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και να διαπραγματευτούμε έτσι ώστε αυτό το Ταμείο Εγγυήσεων να το διαχειρίζεται και τους πόρους να το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε για τον ε, οικονομικό κανονισμό θα συμφωνήσουμε, θα βάλουμε όλα κάτω από το ίδιο ε, καπέλο και να έχουμε με τον τρόπο αυτό την εγγύηση πως ε, θα εγγράφεται στον προπολογισμό και θα το διαχειρίζεται η Κομισιόν με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν, πήγα, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες τώρα για τις διάφορες τροπολογίες, αλλά νομίζω πως εδώ στάθηκα στα θέματα τα οποία θεωρώ πιο σημαντικά. Πολλές τροπολογίες πρέπει απλώς να υπερψηφιστούν γιατί ευθυγραμμίζονται πάρα πολύ με τα όσα εμείς έχουμε υποστηρίξει και αύριο, εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε μία συνεδρίαση με τους σκιώδεις εισηγητές και πρέπει να σου πω ότι προσωπικά έχω συναντηθεί με τους περισσότερους αλλά αύριο έχουμε και μία κοινή συνάντηση για να προσπαθήσουμε να τα καθαρογράψουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική μας θέση και θα περιμένω και εγώ τα δικά σας σχόλια και κυρίως εύχομαι αύριο στη συνάντηση να πάμε με θετικό πνεύμα για να βρούμε το μέγιστο επίπεδο συμφωνίας και να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο έχοντας μια πολύ ισχυρή θέση πίσω μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Συγγήτρια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα όσα είπατε και για την πρότασή σας έτσι ώστε να ξεκινήσουμε με αναπτυξιακή δράση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευχή να καταφέρουμε να επηρεάσουμε την αιτία του προβλήματος. Η κυρία Άουταλα είναι η πρώτη η ομιλήτρια. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι βλέπω κυρία Γουαρδιά Θαμπαλ Ρουβιάλ κατανόησε τις βασικές αρχές του πώς μπορεί να είναι αποτελεσματική η ανάπτυξη οπότε και προσπαθεί να βελτιώσει την πρόταση της Επιτροπής και επομένως να δοθεί ειδικό βάρος στο τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την πολιτική ισότητα των δύο φίλων, οπότε και συμφωνώ επί του προκειμένου με τις προτάσεις της. Ε, επίσης και με τις, ε, το, τις σχετικές τροπολογίες, εκείνες που αφορούν την ε, διαφάνεια, αλλά και την δημοσιοποίηση των φίλων μέτρησης. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με μετανάστευση και ανάπτυξη. Αυτά να μην καλύπτονται από τις ε, νομικές υποχρεώσεις για λόγους νομικούς και πολιτικούς. Βεβαίως και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι προσπάθησε η συντάκτρια να βελτιώσει την πρόταση τη Επιτροπής σε κάποια δύναμα σημεία, αλλά το θέμα είναι κατά πόσον μπορεί κανεί να επιστατεύσει τη σχετική απόφαση για να επισημάνει ε, τις αιτίες της ε, μετανάστευσης. Σε αυτό το σημείο το κείμενο είναι προβληματικό. Δεν νομίζουμε ότι βοηθάει. Όμως, θα μπορούσαμε την πρόταση για να βοηθήσουμε σημαντικά την πολιτική ανάπτυξη της Ένωσης. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτή η παράλληλη πρόταση για το Ταμείο Εγγύσεων θα μπορούσε να είναι ένα μέσο καινοτόμο. Θεωρούμε, επομένως, ότι θα μπορούσε κανείς να κάνει κάτι για την μετανάστευση. Προσοχή να μην διαψευστούν οι προσδοκίες όσων πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όταν μιλούμε για ανάπτυξη, τότε θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ακριβώς τότε ξεκινάει η μετανάστευση, γιατί τότε υπάρχει δυνατότητα μετανάστευσης. Άρα μην θεωρείτε ότι έχουμε στα χέρια μας τη λύση της κρίσης του μεταναστευτικού. Επίσης, νομίζω ότι η προεκοδότηση για την πολιτική που αφορά την αλλαγή του κλίματος είναι πάρα πολύ περιορισμένη, αλλά να πάμε σε άλλη 40% για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την επιτύχηση των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Επίσης, να δούμε τι, τι, τι λέει και για τις ένομες τάξεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Πρόσοχη πώς θα διατεθούν τα χρήματα των φορολογουμένων, εν προκειμένου για κάποια ταμεία που αφορούν κάποια κράτη που δεν συνεργάζονται. Άρα να δούμε εδώ πώς θα δεσμευτούμε όσον αφορά τους επιλέξιμους συνεργάτες μας. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό το άρθρο 11 παράγραφος ένα εδάφιο γάμα που αφορά τους ε, στόχους αναπτυξιακής πολιτικής και ιδίω όσον αφορά το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πώς δηλαδή θα τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα και με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Ευχαριστώ όμω και πάλι την εισηγήτρια και ελπίζω ότι θα αποσπάσουμε αξιόλογα αποτελέσματα κατά αυτόν τον τρόπο. Ο πρόεδρο, εφόσον είναι πάρα πολύ με αυτό το οποίο είπατε, που είναι πολύ θετικά, κύριε Ντεπρέ, για το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δυστυχώ δεν έχω τα χαρτιά μου. Οπότε θα, θα κάνω ό,τι μπορώ. Θέλω να σας πω τα εξή Πρώτα πρώτα όσον αφορά το πρόβλημα της ανακατανομής. Κατά κάποιο τρόπο τίνω να συμφωνήσω με αυτά τα οποία ανέφερε η εισηγήτρια. Άλλωστε τα έχουμε διμερώς συζητήσει. Έχουμε τις ε, τροπολογίες επίσης του ΕΛΚ για την ε, σχέση Ανατολής και Νότου. Θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται για τον Νότο, άρα κατά κάποιο τρόπο να διορθώσουμε αυτά τα οποία προβλέπονται για τις οροφές. Τις οροφές, τα πλαφών της μιας και της άλλης περιοχής. Ε, επίσης είμαι υπέρ του να αυξηθεί το πλαφόν για τη Λατινική Αμερική. Γιατί αν λάβουμε υπόψη το τι ισχύει τι ισχύει για την Λατινική Αμερική, το Μεξικό και την Αμερικανική πολιτική, νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά. Και έτσι θα βελτιωθούν οι σχέσεις με την Λατινική Αμερική. Όμως δεν είμαι υπέρ του να ενταχθεί και η Κούβα στη λίστα αυτή. Και να υποστηρίξουμε έτσι το καθεστώς Κάστρο που δεν έχει προχωρήσει αρκετά όσον αφορά τον αντιδημοκρατισμό. Δεύτερον, όσον αφορά τον στόχο που αφορά άσυλο και μετανάστευση, εδώ υπάρχει το εξή θέμα. Έλαβα υπόψη, όσο είπε η κυρία αλλά και η συγκεντρία. Όμως, από πού και που για να κάνουμε κάτι για τη μετανάστευση μπορούμε κάτι να κάνουμε. Γιατί το, ποια είναι τα προβλήματα, ποιε είναι οι αιτίε. Είναι τα δημογραφικά προβλήματα σε κάποια χώρα. Επίση, οπότε είναι θέμα οικονομική ανάπτυξη. Πού είναι ο στόχο ε, του ότι να υπάρξει ανάπτυξη και απασχόληση για του νέου από αυτέ τι κοινωνίε που έχουν το δημογραφικό πρόβλημα. Οπότε άλλο το σημασιολογικό θέμα και άλλο ο στόχος και η επίτευξή του. Πού είναι οι προοπτικέ ανάπτυξης για να κάνουμε κάτι για τις αιτίε τη μετανάστευσης. Άρα, θα πρέπει να σκεφτούμε ως εξή Πρόεδρε. Όπως και να βλέπουμε τα πράγματα για τις μεταναστευτικές ροές, μεγάλο μέρος της ε, κοινή γνώμης τώρα αισθάνεται πάρα πολύ άβολα γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις ροέ. Άρα πρέπει να δείξει θάρρο η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση αυτών των ροών. Ο κόσμος να μείνει εκεί που να υπάρχει κάποιο είδου ανάπτυξη. Ιδάλω να υπάρχει κάποιο είδους έφτακτη διαχείριση αυτών των ροών στην Ευρώπη. Τώρα όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων, θα πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση, έχουμε κάποιες τροπολογίες, υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις που πολλές φορές είναι υπερβολικές όσον αφορά την ρεαλιστική άποψη των πραγμάτων. Άρα θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Επιτροπής επ' αυτού. Συμφωνώ κατά τα άλλα με όσο είπε η συγγήτρια και θα συζητήσουμε για όλες τις τροπολογίες στην επόμενη συνάντηση αυτές στους τροπολογίες μας βρίσκουν σύμφωνος. Μουρασάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από τη συνάλλητη καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκαρθεθάμπελ για το πολύ επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε, στη συνεργασία της με εμάς και όλες τις συζητητές όπως είπε. Έχουμε αύριο συνάντηση και είμαι αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικέ προτάσει και σε γενική συμφωνία για όλα τα ζητήματα που μας παρουσίασε. Όπως είπε και η ίδια, θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που θα στηρίξει την εισηγήτρια και στις ε, επερχόμενες διαπραγματεύσεις σε σχέση με τα ζητήματα που μας περιέγραψε η εισηγήτρια. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά το γενικό πλαφόν, συμφωνώ με την εισηγήτρια θα ήθελα να υπάρξει αύξηση στα 38,4 δις ευρώ, κάτι το οποίο ευθυγραμμίζεται και με, τις, ε, με τα αιτήματα της ε, ΕΤΕΠ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης θα πρέπει ε, και εμείς να δείξουμε ανάλογο πνεύμα. Σε ό,τι αφορά προκλήσει, υπάρχουν παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις. Θα πρέπει να ιεραρχήσουμε όμως τις προτεραιότητές μας, διότι δεν έχουμε ανεξάντλητους τους πόρους. Ε, είναι πεπερασμένοι και θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε με προσοχή. Και ε, τα προβλήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν προέρχονται από την άμεση γειτονία και ε, την νότια που έχουμε κυρίως στις ζωές μεταναστών και από την ανατολική γειτονία λόγω ε, μιας όλο και πιο επιθετικής τάσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας που φαίνεται να απειλεί κάποιες χώρες ε, της ε, Ανατολικής Γειτονίας που έχουν ξεκινήσει συνεργασία μαζί μας υπό τη μορφή ε, ε, συμφωνιών σύνδεσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε κυρίως ε, στην στηρή εποπτεία βάσει κανόνων και τα ανώτατα ποσά θα πρέπει να δοθούν στην άμεση γειτονία, νότια και ανατολική. Βλέπουμε ότι η Νότια Γετονία λαμβάνει και την ε, ε, μεγαλύτερη υποστήριξη, μεγαλύτερη ενίσχυση μεταξύ των άλλων περιοχών. Η ΕΤΕΠ ε, θεωρεί ότι δεν χρειάζονται επιπλέον πόροι για την Νότια γειτονία. Η εισηγήτρια όμω καταλήγει στο συμπέρασμα πω χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Εμεί είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ω ομάδα αυτή την προσέγγιση. Ωστόσο, δεν θα θέλαμε όλα τα διαθέσιμα περιθώρια να χρησιμοποιηθούν για την νότια γειτονία, διότι θα επηρεαστούν άλλες γειτονίες, κυρίως η Ανατολική. Συμφωνούμε να αυξηθεί ο για τη νοτιά γειτονία, όχι όμως στο ύψος που προτείνει η εισηγήτρια. Είμαστε όμως σε μόνιμη επαφή και ε, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε. Ναι λοιπόν σε αύξηση της νοτιοστονής που ήδη λαμβάνει την υψηλότερη χρηματοδότηση. Το ερώτημα είναι πόσο παραπάνω θα πάρει η νοτιογειτονία ώστε και άλλες περιφέρειες που είναι σημαντικές για εμάς να μην ε, επηρεαστούν αρνητικά. Έρχομαι στην Ανατολική γειτονία. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό η κατάσταση θα έχουμε εξαντλήσει τους πόρους ε, μέχρι το 2018 για την ε, Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και άλλες μικρότερες χώρες. Δεν θα υπάρχει κανένα κονδύλι πλέον. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Έρχομαι στη Λατινική Αμερική. Είναι ώρα να δείξουμε αλληλεγγύη με τη Λατινική Αμερική. Βλέπουμε τις εξελίξεις ΣΥΠΑ που συνιστούν μια σημαντική πρόκληση για τη Λατινική Αμερική και εμείς θα πρέπει να συμπαραταχθούμε με τη Λατινική Αμερική. Η ΕΤΕΠ προτείνει ε, μια κάποια αύξηση για τη Λατινική Αμερική. Είναι αιτιολογημένη, δικαιολογημένη αυτή η αύξηση. Το θέμα είναι το επίπεδο που προτείνει η μπορούμε να το ε, τηρήσουμε, διότι είναι πολύ ψηλότερο από αυτό που προτείνει η, τράπεζα. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να επηρεαστούν αρνητικά οι ενισχύσεις που δίνουμε στην άμεση γειτονία από όπου προέρχονται και βασικές προκλήσεις για εμάς, όπως είπα. Αύριο θα έχουμε συνάντηση με το Σκιώδης, είμαστε σε μόνιμη επαφή ε, με το Γενικό Εισηγητή και θα δούμε όλα αυτά τα πλαφόν που βασίζονται ουσιαστικά στις προτάσεις της ΕΤΕΠ, που αξιολογεί πολύ καλά τις δικές της ανάγκες. Σε ό,τι τους γενικούς στόχους τώρα του Ιελένη. Είμαστε υπέρ της συμπερίληψης συγκεκριμένων στόχων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων στοχευμένων ε, ομάδων μεταναστών, ε, προσφύγων, συγγνώμη. Ξέρουμε ότι έχουν φτάσει πολύ πρόσφυγες τα τελευταία δύο χρόνια στην Ένωση. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φίλων Συμφωνούμε ότι οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην υλοποίηση των έργων όχι όμως κατά τρόπο που θα επιβαρύνει με διοικητικό φόρτο τους τελικούς δικαιούχους. Ό,τι αφορά την σωμάτωση της διάστασης του φίλους πολιτικές, ναι, συμφωνούμε και να εφαρμοστεί όπου είναι εφικτό και δυνατό, αλλά με το σωστό τρόπο. Η συμπερίληψη της Κούβας στις επιλέξιμες χώρες αναφέρθηκε Είναι κάτι που το εξετάσαμε πολύ προσεκτικά ως πολιτική ομάδα οι συνάδελφοί μας, ε, ιδίως από Επιτροπή Άφητα, αλλά και από άλλες επιτροπές, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις. Γνωρίζουμε την περσινή συζήτηση για τη συμπερίληψη της Λευκορωσία ε, στον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών. Ο Ζεράν Ντεπρέ, κατά την άποψή μου, τα είπε πάρα πολύ λογικά. Υπάρχουν σίγουρα θετικές εξελίξεις, μια θετική τάση στις σχέσεις μας με την Κούβα. Όμως δεν είναι τόσο ταχύς ο ρυθμός των αλλαγών στην Κούβα ώστε να την προσθέσουμε στις χώρες τις επιλέξιμες και το θέμα είναι να την προσθέσουμε τώρα ή σε μεταγενέστερο στάδιο ε, με μια κατεξιοδότηση πράξη όπως έκανε η Κομισιόν με τη Λευκορωσία κατά το παρελθόν. Αυτό το θέμα νομίζω θα χρειαστεί να το εξετάσουμε στο επίπεδο των σκιωδών εισηγητών. Επαναλαμβάνω, οι συνάδελφοί μα από την Επιτροπή ΑΦΕΤ έχουν ε, όλο και μεγαλύτερε επιφυλάξει από αυτού. Ταμείο Εγγυήσεων, εν συντομία. Θέλω να πω ότι θα στηρίξουμε την εισηγήτρια. Δεν έχουμε καμία ε, διαφωνία με αυτή τη μεταφορά από ΕΤΕ προς Κομισιόν για να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και σύγκληση με άλλα εργαλεία, με άλλους μηχανισμούς ε, που διαχειρίζεται ήδη η Κομισιόν. Τέλος. Καταθέσαμε μια τροπολογία για αποκλεισμό ε, εξαίρεση μάλλον της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τον κατάλογο των επιλέξιμων χώρων. Γιατί κάνουμε αυτή την πρόταση, διότι βλέπουμε ε, η Ρωσική Ομοσπονδία να έχει όλο και επιθετικότερη στάση απέναντι στην Ένωση και απέναντι σε άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν χορηγεί κονδύλι από το 2014 και μετά επιτόπου. Δεν δίνουμε λοιπόν πιστώσεις, δεν δίνουμε κονδύλια επιτόπου, άρα θα πρέπει αυτό να το ευθυγραμμίσουμε και με τομοθετική μας βάση. Δηλαδή, εισέβαλε σε μια ξένη χώρα η Ρωσική Ομοσπονδία, σε μια χώρα ονόματι Ουκρανία. Έχει προσαρτήσει μια περιοχή ονόματι Κρυμαία. Είναι καιρό πλέον να δώσουμε ένα μήνυμα. Δεν μπορεί να συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, ε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα σε ό,τι δεν αφορά τη σχέση μεταξύ Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θέλουμε να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα Εγώ νομίζω ότι η νομοθετική βάση πρέπει να ευθυγραμμιστεί με αυτή την πραγματικότητα επιτόπου, δηλαδή δεν χορηγούνται πλέον κονδύλια στην Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά από πλευρά μου και θα συνεργαστούμε με τα χαρά την εισηγήτρια, του κοιόδε εισηγητέ, ε, του υπόλοιπου, ώστε να καταλήξουμε σε ευρεία συνένεση και να έχουμε μια πιστική πλειοψηφία από πλευρά Κοινοβουλίου για τι επερχόμενε διαπραγματεύσει. σα ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Κιόλμελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Είναι πολύ ε, διεξοδική η δουλειά της και στηρίζουμε ως ομάδα τα περισσότερα στοιχεία αυτής της έκθεσης. Θέλω να συγχαρώ επίσης ε, τους ε, νεοεκλεγέντες αντιπροέδρους και την εκλεγής αντιπροέδρα. Τώρα, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για το κατά πόσο να αυτό το οποίο προτείνουμε εδώ ε, στην Επιτροπή μας ε, είναι ε, από πλευράς τακτικής ευφυές και σωστό. Και σε ό,τι αφορά το τίτλο για αυτήν την έκθεση, δηλαδή τα μεγκύσω για τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπάρχουν και θέματα αναπτυξιακής βοήθειας, στήριξης ε, της δημοκρατικής ε, ανάπτυξης ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά τελικά υπάρχουν και πολλές αλλαγές, πολλές τροπολογίες με τις οποίες θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεταναστευτική κρίση. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Θέλουμε να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, αλλά θα πρέπει να είναι διαφορετικό αυτό το μήνυμα με μια έκθεση που αναφέρουμε κάποια νούμερα, ε, δεν νομίζω ότι αρκεί αυτό και δεν είναι αυτή η διαφάνεια που αναμένουν από εμάς οι πολίτες. Πρέπει, ίσως να το κάνουμε και αυτό, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε και μια άλλη προσέγγιση ό,τι αφορά τη μεταναστευτική κρίση. Θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε στα, ε, στις ρίζες, στα βασικά της αίτια, με αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε αν μέσω ενός ταμείου εγγυήσεων θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεταναστευτική κρίση, γιατί αυτό στην πράξη τι θα σήμαινε. Θα σήμαινε ότι εμείς ως Κοινοβούλιο ουσιαστικά θα έχουμε ε, λίγες δυνατότητες ε, σε ό,τι αφορά ε, τις επενδυτικές δράσεις. Το πώς θα μπορούμε να αναλάβουμε τη διαχείριση σε ό,τι αφορά την ΕΤΕΠ, την οποία την εμπιστεύομαι βέβαια, δεν ξέρουμε στην πράξη τι γίνεται. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα ως προς αυτό. Επίσης ξεκάθαρα θα πρέπει να είναι το ότι ενδεχομένως ε, θα έχουμε ασκήσει μια ε, πολιτική αναπτυξιακή που ε, κατά το παρελθόν απεδείχθη ανεπαρκής και εσφαλμένη σε ό,τι αφορά τις δομές. Δεν ενισχύθηκαν τελικά. Δημιουργήθηκαν νέες δομές και υποβαθμίστηκαν οι δομές υφιστάμενες. Αυτό θα μπορούσε να ξανασυμβεί και θα μπορούσε να υπάρξει και ε, πρόβλημα με τον ανταγωνισμό. Θέλουμε σίγουρα να επενδύσουμε ε, με ασφαλή δάνεια από την ΕΤΕΠ. Το θέμα είναι όμως πώς όλα αυτά θα επηρεάσουν τον ανταγωνισμό. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα λοιπόν. Άμεσες επενδύσεις Ευρωπαϊκή Ένωσης. Νομίζω αυτό ε, θα μας δώσει τη δυνατότητα να περάσουμε περισσότερο και να εστιάσουμε σε τομείς που δεν θα βλάψουν τις εγχώριες οικονομίες, περιβάλλον, προστασία περιβάλλοντο για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να επενδύσουμε επίσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης. Δεν βλέπω προβλήματα εκεί ε, για την εγχώρια οικονομία, αλλά ε, θα πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα και να πούμε ξεκάθαρα πόσα χρήματα θα κοστίσει αυτό, πόσα χρήματα αξίζει να δοθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ υποστηρίζω εδώ και καιρό ε, ότι θα πρέπει να δώσουμε χρήματα, πολλά χρήματα ε, σε αυτό το τομέα θα ήταν κάτι θετικό, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε ένα συνολικό κόνσεπτ, ε, μια συνολική αντίληψη για την μετανάστευση και το προσφυγικό αλλιώς θα είναι μόνο μερική η προσέγγιση και η αντιμετώπιση. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα για να πετύχουμε τους στόχους. Επομένω, συνολικά θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η δουλειά της εισηγήτρια σε ό,τι αφορά τον τομέα της αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης ε, εισαγωγικά, εντό εισαγωγικών να μην την πνίξουμε, να μην την περιορίσουμε σε μια τέτοια έκθεση, αλλά να δούμε σημαντικά ουσιαστικά τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον Μπενίτο Σιρουάδα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μόνο κάποια γενικά σχόλια για τις εκθέσεις τις οποίες συζητάμε εδώ για τη χρηματοδότηση εξωτερικής δράσης της ΕΤΕ. Για πάρα πολλά χρόνια η... το θεματολόγιο για την ανάπτυξη των φτωχοποιημένων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν ένα θέμα για μας δευτερεύον και νομίζω ότι είναι μεγάλη σύμπτωση το γεγονός ότι τώρα α, κοιτάμε τι γίνεται με την ανάπτυξη στις τρίτες χώρες ε, σε μια χρονική στιγμή που συμπίπτει με το προσφυγικό. Νομίζω ότι είναι αποφάσεις οποίες πιεστήκαμε να πάρουμε και νομίζω ότι έτσι θέλουμε να καλύψουμε τις ανησυχίες των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν επειδή υπάρχει αυτή η σύμπτωση με την κρίση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιορισμένων δημόσιων πόρων που χρησιμοποιήθηκαν, είπαμε να χρησιμοποιήσουμε ε, χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Εύση, όπως επίσης και κάποια άλλη μηχανισμοί, ιδιωτικές επενδύσεις, ΣΔΙΤ, δημόσιες επενδύσεις, ε, και αυτό λόγω των χαμηλών αποδόσεων που έχουν αυτές οι δράσεις αν επενδυθούν ε, μόνο ιδιωτικά ε, κεφάλαια. Έτσι λοιπόν η απόφαση αυτή θέλει να στηρίξει και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί έτσι ώστε οι επενδυτές αυτοί, οι ιδιώτες επενδυτές να έχουν μειωμένους κινδύνους με την ελπίδα πως οι χώρες που θα επιλεχθούν θα καταφέρουν τελικά να δεχτούν τους μετανάστες που επιστρέφουμε από τις χώρες μας Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά κάποια εδάφη τα οποία θα περιορίζουν τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας και θα δώσουμε αυτό και κάποιες ευκαιρίες ε, ε επιχειρηματικής δράσης σε ευρωπαϊκές εταιρείες ή ολιγάρχες της περιοχής. Άρα λοιπόν πρέπει να σας πω πως στις χώρες αυτές το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τις άμεσες επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με ανταλλαγές δίκαιες και συνεργατικές, ε, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή ε, και πιστεύω πως τα σχέδια αυτά ε, των επενδύσεων που έχουμε αντικατοπτρίζουν τα όσα σας περιγράφω. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε υπέρ της στήριξης τέτοιου είδους χρηματοδότησης. Merci. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκράσλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επισώ την προσοχή σας στο ότι ε, σε ό,τι αφορά αυτό ε, το δορυφορικό δημοσιονομικό σύστημα, όπως το λέμε, για το οποίο αρκετές φορές έχουμε εκφράσει τη δυσαρέσκειά μας ε, σε ό,τι αφορά αυτό το δορυφορικό σύστημα. Έξι δις ε, είναι το ποσό το συμπληρωματικό που θέλουμε να δώσουμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι εντελώ ασυνεπέ σε ό,τι δεν αφορά την πρώτη πρόταση τη εισηγήτρια. Νομίζω ότι με την πρόταση τη Κομισιόν ε, πρέπει να προχωρήσουμε, όχι να διευρύνουμε την προκοδότηση του Ταμείου Εγγυησέων και στην πρόταση της Κομισιόν και στι δικέ μα ε, προτάσει σε ό,τι αφορά αυτό το Ταμείο Εγγυήσεων θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα άλλα προγράμματα και τις πολιτικές. Έχουμε την πολιτική γειτονία 18 ε, δις για, την, ε, για τον τομέα αυτό. Όμως βλέπουμε ότι δεν, ρέει, δεν ρέουν τα χρήματα αυτά στα προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, δούμε τι θα κάνουμε και σε ό,τι αφορά ε, και αυτό που λέει η Κομισιόν ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση να συνδέεται και με την δυνατότητα απορρόφησης και εκτέλεσης. Επομένως δεν νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε γιατί δεν υπάρχει σύνδεση μέχρι στιγμή, με τα μέχρι στιγμής προγράμματα. υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού μεταξύ των προγραμμάτων της Ένωσης και της ΕΤΕΠ. Το πρόβλημα είναι και η περιορισμένη δυνατότητα διαχείρισης αυτών των προγραμμάτων επιτόπου. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί. Ένα δεύτερο ε, ή μάλλον τρίτο ερώτημα για τα έξι δις, ε, τα επιπλέον ε, είπα ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτό το τομέα γιατί να τα δώσουμε αυτά τα χρήματα. Δεύτερο ήταν αυτή η σύνδεση που είπαμε τα ευστάμενα προγράμματα και τρίτο θέμα Λατινική Αμερική που παίρνει 5 δις Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την μετανάστευση. Δεν είδα να έρχονται και τόσοι πια μετανάστες από την Λατινική Αμερική. Έχει νόημα λοιπόν για τη Λατινική Αμερική. που οι Αμερικάνοι φίλοι μας ε, ε, έχουν εκφράσει τη δική τους ε, ευθύνη εντό αγωγικών για αυτήν την περιοχή, γιατί εμείς να αναλάβουμε να βοηθήσουμε με τόσο μεγάλα ποσά, το θεωρώ και αυτό μη συνεκτικό ως πρόταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάουταλα πάλι μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πατήσω σε κάποια από τα σχόλια που άκουσα. Κύριε Ντεπρέ, αντιμετωπίσατε με σκεπτικισμό τα σχόλιά μας. για την αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν τη μετανάστευση. Αλλά η ερώτηση δική μου είναι γιατί εμείς θα πρέπει να εφεύρουμε εκ νέου τον τροχό. Έχουμε πολύ ε, καλές αρχές πάνω στην οποία βασίζουν την απτυξιακή πολιτική και τώρα ε, που ξεκινήσαμε γιατί να μην τα βάλουμε όλα ε, κάτω από την ομπρέλα αυτή. Νομίζω πως αν μιλήσουμε μόνο ε, για τις γενεσιουργές αιτίε, τότε δημιουργούμε σύγχυση με τις αρχές που ακολουθούμε στην αναπτυξιακή πολιτική. Και γι' αυτό ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια τροπολογία της εισηγήτριας που ε, προκαλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει έναν ε, κατάλογο με τις γενεσιουργές αιτίε τη μετανάστευση, που νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να το κάνει. Καταλαβαίνω όμως γιατί το ζητάει η εισηγήτρια μάλλον. Κύριε Κέλμελ, δεν νομίζω πως η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποτύχει. Νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε πιο κοντά στις αρχές της, να δημιουργήσουμε περισσότερους μηχανισμούς εποπτείας, λογοδοσίας, διαφάνειας, παρακολούθησης και βέβαια το κάνουμε νομίζω πως ε, θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη σύγχυση ιδεών που προκαλεί η αναφορά στην ουσιοργία τη μετανάστευση. Και αν το κάνουμε, δεν νομίζουμε ότι για την αναπτυξιακή πολιτική μα και τι αρχέ που τη διέπουν, αυτό είναι σωστό. Τώρα, για το Ταμείο Αγγίσεων. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε, να στήσουμε ένα σύγχρονο εργαλείο που θα προσκαλέσει τον ιδιωτικό κλάδο να συνεισφέρει στους αναπτυξιακούς μας στόχους και σε πιο δύσκολες χώρες και σε έθραυστα κράτη. Ίσως είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι, αλλά αυτό είναι η βασική έννοια. Θα πρέπει τα χρήματα των φορολογούμενων να μοχλεύσουν ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία δημιουργούν αναπτυξιακά παραδοτέα. Και γι' αυτό οι σκιώδεις εξετάζουν με... και παρακολουθούν στενά τη βασική ε, πρόταση που έχει να κάνει με το Ταμείο για την ε, βιώσιμη αναπτυξιακή βοήθεια. Η Μπιελορούς, η Λευκορωσία, θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για τα κονδύλια τα οποία συζητάμε. Και η Ρωσία όχι. Merci. Σας ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν. Θα ζητήσω τώρα από την εισηγήτρια να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν θέσει οι συνάδελφοι, οι οποίοι πήραν το λόγο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και σε επικοινωνιακό επίπεδο ή θα θεωρηθεί πως είναι ένα εργαλείο για να καταπολεμήσουμε τη μετανάστευση που δημιουργεί προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι λοιπόν μια επικοινωνία με τους συμπολίτε μας για να κατανοήσουν το εύρος και την συνοχή που υπάρχει στις πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να μας διευκρινίσετε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό, τι θα συμβεί με τις εγγυήσεις άμα περάσουμε στα 36 δις. Θα πρέπει ως εγγύηση λοιπόν να εγγράψουμε κάποιο ποσό στον προπολογισμό να δούμε πώς αυτά όλα θα χρηματοδοτηθούν. Έχετε το λόγο συνάδελφε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αν όχι σε όλους, τουλάχιστον να σας πω κάποιες σκέψεις μου και πρώτα-πρώτα για κάτι που μας απασχόλησαν πάρα πολύ όσον αφορά τους νέους ε, στόχους και την καταπολέμηση των ε, ριζών της μετανάστευσης των αιτίων. Ε, είπατε κύριε Ντεπρέ ότι είναι και θέμα σημασιολογικό ε, ναι, πρόκειται περί τούτου, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιούμε κάποια φρασιολογία και όχι άλλη και υπάρχει λόγος για την επιλογή μας αυτή και νομίζω ότι παρά το ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο κατά να προσπαθούμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη από τη μια και από την άλλη να θέλουμε να κάνουμε κάτι για τη μετανάστευση. Το ένα μου φαίνεται ε, πιο, πιο δυναμικό. Το άλλο μου φαίνεται ε, κάτι πιο αρνητικό εντός ε, εισαγωγικών και δεν συμφωνώ με, αυτό το δεύτερο. Άρα το θέμα είναι το τι φασουλία χρησιμοποιούμε που μας οδηγεί και στο τι κάνουμε για το πρόβλημα. Οπότε ανεξάρτητα από το τι διατύπωση θα χρησιμοποιήσουμε, ε, αν θα μιλήσουμε δηλαδή για αιτίες ε, μετανάστευσης ε, ή για αιτίες της ε, μετανάστευσης. Έχει τρεις στόχους είπαμε, η ΕΤΕ, δηλαδή το, πώς θα αναπτύξουμε τον ιδιωτικό τομέα για τις ΜΜΕ στις χώρες εκείνες, τι θα γίνει με τις υποδομές, με μεταφορές, ενέργεια, πολιτικές περιβάλλοντος, τηλεπικοινωνίες και αλλαγή του κλίματος. Γι' αυτό το, το, το λέμε ως γενική σκέψη, χωρίς να μπούμε στις λεπτομέρειες. Έχουμε στην Ευρώπη και βέβαια στην Ισπανία πολλούς μετανάστες από την Λατινική Αμερική, αλλά δεν αναφέρεται εδώ ούτε η μετανάστευση από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες, αλλά στη Λατινική Αμερική βέβαια έχει πολλές μεταναστευτικές ροές, οπότε αυτό θα πρέπει να δούμε το ότι στις χώρες εκείνες έχει, έχει ο κόσμος τη ζωή του και δεν θέλει να μετακινηθεί. Οπότε υπάρχει και ένας στόχος πολύ πιο γενικότερος. Μισό ότι έχω πολλά σημειώσει εδώ, μην ξεχάσω τίποτα. Τώρα, γι' αυτό που είπε η κυρία Χάουταλα, δηλαδή να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει τις αιτίες της ε, μετανάστευσης και είπαμε ότι θα πρέπει τις ε, απότερες αιτίες να τις ε, αντιμετωπίσουμε, root causes, λέει, για να δούμε κατά πόσον τα μέσα πολιτικής που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι τα πιο δόκιμα για να μπορέσουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουν. Οπότε ε, συμφωνούμε και να υπάρχει αυτό στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε να στοθούμε στη δουλειά και να δούμε ποια είναι τα αναγκαία εργαλεία προς Κυρία Γκρέσλε μας είπε ε, για το δορυφορικό σύστημα και η αύξηση της εγγύησης είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι θέμα ποσοτικής αύξησης και αυτό θα έχει συνέπειε στον προπολογισμό. Σύμφωνα με το σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο χρειαζόμαστε 35 εκατομμύρια. Αυτό είναι το θαύμα, είναι σαν τους άρτους και τα ψάρια στην βίβλο. Τι θα κάνουμε με τα 35 εκατομμύρια, πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αύξηση της συνολικής εγγύησης. 35 εκατομμύρια όντως φτάνουν μέχρι το 2020 Οπότε υπάρχει και αυτή η δέσμευση για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πώς θα γίνει τώρα να δώσουμε το πράσινο φως, όχι επισήμως, αλλά έχει γίνει αυτό και θα έχουμε δεδομένη την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου. Οπότε το συνολικό περιθώριο για τις υποχρεώσεις μας αυτό θα είναι και θα υπάρχει και ασφάλεια. Το 3 δεν είναι τίποτα το, το δύσκολο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ωραία, θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούμε αύριο πρωί. Ευχαριστώ κύριε Γκουρθάπολ. Τώρα κάτι τεχνικής φύσεως. Η εγγύηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αφορά το σύνολο του δανείου λέει ο πρόεδρος. Δηλαδή, εάν δεν είσαι κανείς ένα δις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει εγγύηση στην Τράπεζα Επενδύσεων. Και εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο, εάν φτωχεύσει ε, ο, ο φιλέτης, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον υποκαθιστά. Και τι ποσοστό καλύπτει αυτή η εγγύηση, σε τι ποσοστό ανέρχεται μάλλον, 65% του δανείου. Υπάρχει εκπρόσωπος της Τράπεζας Επενδύσεων. Μπορείτε να μας απαντήσετε από αυτού. Εάν κανείς δανείσει 100, πόσο είναι η εγγύηση από τον προηγούμενο της Ένωσης, και απαξί συμφωνηθεί το δάνειο τι πρέπει να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν εγγύηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να, το, να σας απαντήσω όπως και συνάδελφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 65% με πληρωμές 9% ε, από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9% de 65%. το 65% δηλαδή να καταλάβω. Δηλαδή 6 δις επιπλέον, 4 δις είναι τα 65%, 65% και 9% το 4 δις 360 εκατομμύρια που θα πρέπει να εγγραφούν από, στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά, 9% λοιπόν του 65% από τον προπολογισμό. Δηλαδή αυτό μην το ξεχνάτε. Pour la Commission, Monsieur Angel. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να σας απαντήσω, η απάντηση δεν ήταν ακριβώς, ε, δεν έγινε ακριβώς κατανοητή. Το 9% είναι για την ολόκληρη διάρκεια της εγγύησης. Δηλαδή, αν δώσουμε 38 δις, όπως θέλει να το κάνει, θα πρέπει να έχουμε 9% του 38,4 δις. Τώρα, ο όγκος της εγγύησης, εκτός ε, μικροφώνου πρόεδρος, Δυστυχώς είναι εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Το σύνολο της εγγύησης, δηλαδή δίνουμε μια εγγύηση στο 100% αλλά με περιορισμό που να είναι τουλάχιστον το 65% του ολόκληρου χαρτοφυλακίου. Δεν είναι δηλαδή ένα project, είναι εγγύηση για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των project που είναι τουλάχιστον 65%. Αν λοιπόν επιλέξετε λοιπόν, να έχετε αυτό το 38,4 δις που είναι υψηλότερο από αυτό το οποίο είχαν διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, de facto μέγιστος κίνδυνος για το ευρωπαϊκό προβλήμα είναι 65% αυτού του ποσού, αλλά για συγκεκριμένο project, όσο δεν έχουμε φτάσει το 65%, μπορεί να είναι και το 100%. Ελπίζω να ήμουν σαφής, είναι λίγο θα ήθελα να επιμείνω εδώ, δηλαδή η δημοσιονομική επίπτωση μιας τέτοιας απόφασης είναι στα, στις δαπάνες να εντάξουμε τα απαραίτητα κονδύλια για την κατάθεση της εγγύησης που είναι το 90% των 36 δις. Αν αυξήσουμε κατά 6 δις θα πρέπει από αυτά τα 6 δις να βρούμε άλλα 9% για τον προϋπολογισμό μας. Δηλαδή 540 εκατομμύρια ουσιαστικά. Θα μείνουμε εκεί. Σας ευχαριστώ. Πολύ σημαντική η αυριανή συνάντηση. 27 Μαρτίου, σε έξι μέρες μπορούμε να εγκρίνουμε την έκθεση. Εντολή 1η Απριλίου και πρώτος τριμερής διάλογος 10 Απριλίου. Προς επιβεβαίωση βέβαια η ημερομηνία. Ευχαριστώ την εισηγήτρια θα δώσω μετά το λόγο στον επόμενο εισηγητή ε, μακροοικονομική βοήθεια στην Μολδαβία, ο κύριος Μούρεσαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά απλή διαδικασία. Γι' αυτό και έχουμε πολύ λίγη ε, ώρα για τη συζήτηση. Στον Ιανουάριο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ στην ε, Δημοκρατία τη Μολδαβία ω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή για να στηριχθεί η μικρή αυτή χώρα τη Ανατολική Γειτονία ε, τα οποία χρήματα αυτά θα πρέπει να δοθούν ως 40 εκατομμύρια ως ε, επιχορηγήσεις και 60 ως πιστώσεις σε μια περίοδο 2,5 ετών με δόσεις. Και βέβαια πάντοτε θα πρέπει να τηρείται αυστηρά το μνημόνιο συνενώσεις που θα συμφωνηθεί και θα υπογραφεί από Ευρωπαϊκή Υποτροπή και Δημοκρατία της Μολδαβίας. Αυτά ήταν τα αρχικά. Πού βρισκόμαστε τώρα και ποια είναι η δική μου άποψη για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, εφόσον καθήλυνα αρμόδια είναι Επιτροπή ΙΝΤΑ. Εμείς γνωμοδοτούμε απλά. Υπάρχουν αρκετέ προποθέσει βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δίνει ε, πιστό στη ε, δημοκρατία τη Μολδαβία μόνο εάν πληρούνται τα δημοκρατικά πρότυπα, να σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν υπάρχει κράτο δικαίου. Αυτέ οι προποθέσει φυσικά είναι γενικέ. Δεν μπορούμε να τι αλλάξουμε. Και πιστεύω ότι οι προποθέσει αυτέ, ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου, τηρούνται. Άρα μπορούμε να περάσουμε πλέον στο επόμενο στάδιο που είναι συζήτηση ενός πολύ συγκεκριμένου μνημονίου ε, κατανοές συμφωνίας ε, που θα αποφασιστεί και θα ψηφιστεί από, θα υπογραφεί τέλος πάντων από την Κομισιόν και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας όπως είπα. Αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο με σαφείς απτούς στόχους και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα πρέπει να τα επιτελέσει η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η κυβέρνηση της Μολδαβίας, να ενισχύσει περισσότερο το δικαστικό σώμα, καταπολέμηση της διαφθοράς, ένας άλλος στόχος, η ε, υποστήριξη της όλο μεγαλύτερη ανεξαρτησίας ε, των δικαστών, εισαγγελέων, ε, αντιμετώπιση ξεπλήματο χρήματο, ενίσχυση του τραπεζικού τομέα, μεγάλη τραπεζική απάτη το 2014 στη Μολδαβία 1,1 δις ευρώ πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα. Έτσι προτείνω να προχωρήσουμε με την έκθεση να δετεθούν τα χρήματα για τη χώρα αυτή, όπως προτείνει η Κομισιόν, όμως στο μνημόνιο αυτό ε, συμφωνία μεταξύ Κομισιόν και Δημοκρατία της Μολδαβία, επιμένουμε να αναφέρονται συγκεκριμένοι όροι. Και αυτά τα πιο συγκεκριμένα θα τα δείτε στις τροπολογίες. Σαφείς ώρες, λοιπόν και προποθέσει. Αυτό περιμένει και ο λαός της χώρας. Να είμαστε στο πλευρό του περιμένει. Γενικά να στηρίζουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. αλλά αν χρησιμοποιούμε του περιορισμένους οικονομικούς πόρους που έχει η Ένωση σωστά, αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει οι χώρε για τι οποίε ε, παρέχουμε βοήθεια να βελτιώνονται. Και σίγουρα και για τη Μολδαβία ισχύει αυτό. Υπάρχει συμφωνία σύνδεση με την Ένωση, άρα είναι ισχυρή η σχέση μα. Θα πρέπει η χώρα να παραμείνει ε, στο δρόμο των ε, μεταρρυθμίσεων, να εφαρμόσει και τα συμπεφωνημένα στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης. Ε. Αυτή θα είναι λοιπόν η γραμμή των τροπολογιών που θα καταθέσω. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών κύριε Πρόεδρε, η 23η Μαρτίου, 10 το πρωί. Η ψηφοφορία για την έκθεση ε, προβλέπεται στην Επιτροπή μας για τις 3 Απριλίου, για να μπορέσουμε λοιπόν να αποχωρήσουμε αυτό το μνημόνιο και να διατεθούν τα χρήματα στην Μολδαβία. Πάντα, όπως είπα βέβαια, βάσει σαφών μετρήσιμων όρων και προποθέσεων. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. φύγει τα όσα μας είπε το κύριο Νεγκρέσκου. Ευχαριστώ. Επειδή θα φτάσει ε, το μήνυμά μου και στη Δημοκρατία της ε, Μολδαβίας ε, και θέλω να με καταλάβω, θέλω να πω ότι αυτή η έκθεση δείχνει το ανοιχτό πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Δημοκρατία της Μολδαβίας και λαμβάνει υπόψη όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχουν επιτελεστεί εκεί. Δεν θα πρέπει να έχει πολιτική χρειά η έκθεση. Θα πρέπει να αναλύσουμε αυστηρά δημοσιονομικά ε, τα διάφορα στοιχεία. σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το πνεύμα της Επιτροπής ΙΝΤΑ και εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν πιο απλοί και συγκεκριμένοι. Δεν θα πάνε στην κυβέρνηση τα κονδύλια αυτά, αλλά στο λαό της χώρας και έχουμε τις προϋποθέσεις ε, τη συνήθως προστασία ε, κράτος δικαίου, ε, δημοκρατία, πολέμηση διαφθάση κτλ. κτλ. Θα πρέπει να είναι λοιπόν μια ασφαλιστική δικλίδα αυτές οι προϋποθέσεις για να πάνε τα χρήματα στο λαό δηλαδή ιδίως στο σημερινό πλαίσιο. Πρέπει να δείξουμε πόσο στηρίζουμε τη Μολδαβία. Ελπίζω να μην πολιτικοποιηθεί έκθεση και να παραμείνει σε αυστηρά δημοσιονομικά πλαίσια. Πρόεδρος. Ποια άλλη θέλουν το λόγο, ε, γιατί δεν θέλω να άνοιξω κατάλογο. Κύριο Στάρεν ήταν τελευταίο. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω πως γενικά συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητή. Ο κύριος Νεγκρέσου καθώς με προκάλεσε και θα πάρω το λόγο. για να μην περιορίσουμε την έκθεση αυτή μόνο σε δημοσιονομικά θέματα. Αυτό μου δημιουργεί κάποια προβλήματα, γιατί γνωρίζετε κι εσείς πως οι τράπεζες στη Μολδαβία εμπλέκονται, δυστυχώς, ε, με άλλες, ε, με άλλες τράπεζες δυστυχώς ιστονικές, λιθουανικές, ε, λετονικές και ε, δανέζικες σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε η κυβέρνηση Μολδαβίας, αγαπητέ συνάδελφε, να χρησιμοποιήσει τη συμφωνία Eurojust για παράδειγμα για να ερευνήσει το θέμα, για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση στο θέμα αυτό, για να αποφεύγονται τέτοιου είδες πρακτικές. Και μια τελευταία πρόταση. Πραγματικά πιστεύω πολύ στους Μολδαβούς ε, στρατιώτες, τους οποίους το 1983 εγώ δίδασκα ε, στο Σοβιετικό στρατό. Πολύ καλοί στρατιώτες, αλλά εξαιρετικοί και στον δωροδοκούν όταν ήθελαν μετάθεση σε κάποια πόλη, μου έφερναν οι γονεί του κρασιά για να μετατεθούν. Οπότε καταλαβαίνετε πώ ε, η κατάσταση εδώ είναι ε, σοβαρή και θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Euh, νομίζω πως ο εισηγητής έχει ένα κείμενο εδώ ξεκάθαρο για το σημείο. Αν δεν ζητάει κάποιο άλλο το λόγο, νομίζω ότι αγαπητέ εισηγητή μπορούμε να μείνουμε εδώ και θα το ψηφίσουμε 3 Απριλίου. Θα δώσω το λόγο τώρα στο αδελφό κύριο Νεγκρέσκο για το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ έχουμε μια γνωμοδότηση για την τεχνική βοήθεια και εδώ πρόκειται για πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μιλήσω αγγλικά. Δεν έχω πολλά σχόλια να κάνω. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί στην τεχνική βοήθεια να κατανείμει κάποια ποσά. Ξέρετε πώς θα μπορούσε να πάει στο 0,5 του σχετικού προπολογισμού του Ταμείου. Φέτος θα μειωθεί από τις 380.000 ευρώ στις 310.000 ευρώ, το οποίο σημαίνει 0,18% του συνολικού προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια πρόταση και υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσφοράς ε, τεχνικής βοήθειας, καλύτερη εποπτεία και συλλογή δεδομένων και εργαλεία σχετικά, Έχουμε για παράδειγμα την ανταλλαγή των πληροφοριών, με την οργάνωση δύο συναντήσεων εμπειρογνωμόνων. Όλα μοιάζουν σωστά, ενδιαφέροντα. Η δική μου διάσταση που προσθέτω στην έκθεση και ελπίζω θα με βοηθήσετε, γιατί έχουμε συζητήσει το Ταμείο αυτό πολύ συχνά, είναι πρώτα απ' όλα θα πρέπει η επικοινωνία ε, με τις ευκαιρίες που δίνει το Ταμείο αυτό να, και με τους ευνο, ε, ωφελούμενους και τους δικαιούχους να βελτιωθούν. Επίσης, βέλτιστες πρακτικές, αυτό δεν αναφέρεται στην πρόταση της Κομισιόν, θα πρέπει να είναι πιο ενεργητική στην εμπλοκή των εθνικών σημείων επαφής. Κάποια κάνουν καλά τη δουλειά τους, κάποια όχι. Οπότε θα πρέπει να εντοπίσουμε τους χώρους στους οποίους χρειάζεται να κάνουμε προσπάθεια και να ζητήσουμε τα εθνικά σημεία επαφή να αναλάβουν μεγαλύτερη δράση. Και τέλος, αλλά όχι ίσονος σημασία, η έκθεση αυτή μιλά για μία ε, ένα επιπρόσθετο στοιχείο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ε, Παγκοσμιοποίησης που πρόσθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το κριτήριο της κινητοποίησης λόγω κρίσης που θα ευξήσει κατά 60% την ε, χρηματοδότηση και θα βοηθήσει να διαχειρίζεται πιο εύκολα τους φακέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέροντα αυτά λοιπόν στην έκθεση, ήθελα να τα υπογραμμίσω και να σας πω ότι προέρχεται από εμά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν είναι καλό. Ευχαριστώ και πρέπει να αναφερθεί. Merci. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Σιγητάλη ο Πρόεδρος. Ζητεί κάποιος το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Πάντως μου φαίνεται κάποιος θλιβερό ότι ενεργοποιείται το Ταμείο μόνο κατόπιν των απολύσεων. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο τρόπο να βοηθούν οι επιχείρησει που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Οι τροπολογίε πρέπει να καταδεχθούν πριν στις 27 Μαρτίου το μεσημέρι, ημέρα Δευτέρα. 3 Απριλίου στην Επιτροπή θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια θα ψηφιστεί ε, στις 4 Απριλίου. Ο κύριος Ντεπρέτορα έχει το λόγο για την μετεγκατάσταση των ε, μεταναστών και των άσυλων και προσφύγων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να είμαι πολύ σύντομος, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω τροπολογίες από πλευράς της Επιτροπής των Προϋπολογιστών για αυτό το σημαντικό πρόγραμμα πλαίσιο. Να δούμε τώρα τα δημοσιονομικά. Πρώτα πρώτα να γίνει κάποια διάκριση, συνάδελφε, μεταξύ της ε, μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης. Αφορά κάποιους που βρίσκονται σε κάποιους ατόμπε, ας πούμε, στην ε, Περιορδανία, στη Συρία, Ιράκ και Τουρκία και τότε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους δέχονται στην επικρατεία τους. Αυτό είναι η μετεγκατάσταση και περί τούτου πρόκειται. Ε, προκειμένου η επανεγκατάσταση είναι αυτό το οποίο προβλέπεται από την μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών από πλευράς προϋπολογισμού είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε το τι θα πρέπει να προβλέπετε στους επόμενους προπολογισμού, μια που θα πρέπει η Επιτροπή κάθε χρόνο να διατυπώσει πρόταση για το πόσοι πρόκειται να μετεγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τα κράτη-μέλη όμως έχουν αρμοδιότητα να πούν το πόσους δέχονται. Άρα δεν έχουμε τη βάση υπολογισμού του πιθανού κόστους μιας τέτοιας κίνησης. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο ρητός προβλέπεται εν προκειμένου, το οποίο επιβιώνει τη σημερινή πρακτική, είναι ότι κάθε κράτος μέλος το οποίο δέχεται ε, να εγκατασταθεί κάποιος, πρόκειται να υποστηριχθεί από τον προπολογισμό και ε, από το Ταμείο ΑΜΙΦ το ποσό των 10.000 ευρώ. Αυτό ήδη προβλέπεται, δεν είναι καινούργιο. Όμω, από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο είναι μια καινοτομία και με βρίσκει σύμφωνο, είναι το ότι μέχρι σήμερα, όταν τα κράτη-μέλη αποφασίζουν πέραν του ευρωπαϊκού πλαισίου με την κατάσταση το οποίο συζητούμε τώρα, εάν α πούμε διμερό έχουν συμφωνήσει να εγκαταθούν κάποιοι στην επικρατειά του, πρόκειται να έχουν 6.000 ευρώ από τον κοινωνικό προπολογισμό. Και εγώ θεωρώ ότι Αφού θέλουμε να έχουμε ένα ενωσιακό πλαίσιο για την μετεγκατάσταση, τότε είναι φυσιολογικό να παρέμβει για τη χρηματοδότηση ο προπολογισμό για τα πρόσωπα αυτά που θα μετεγκατασταθούν. Από την άλλη μεριά. Από πού και ως πού, με βάση ποια επιχειρήματα θα συνεχίσει ο προπολογισμό να επιδοτεί, να ενισχύει τις χώρες που αποφασίζουν να μετεγκατασταθούν κάποιοι στην επικρατειά τους πέραν του ενωσιακού πλαισίου. Οπότε συμφωνώ με αυτές τις δύο προτάσεις που διατυπώνονται στο έγγραφο το οποίο έχετε λάβει και το συζητούμενο έγγραφο και δεν έχω κάποιες τροπολογίες από πλευράς δημοσιονομικής για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχω τροπολογίες αλλά αυτό είναι άλλο παπαγγελία. Ευχαριστούμε κύριε ο πρόεδρος. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Κύριε Γιώτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του και συμφωνώ. Και δεν έχω και πολλά να προσθέσω στα όσα είπε ο εισηγητής Ντεπρέα. Σύμφωνα με το πνεύμα που διαπνέει το κείμενό του και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η δουλειά και από πλευρά Επιτροπή των Προπολογισμών. Σε σχέση με τον στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Και πάλι μπράβο στον συνάδελφο για τη δουλειά του. Ευχαριστούμε. Κύριε Σαρβαμά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, uh, Βέβαια. Βέβαια και χρειαζόμαστε. Να, αυτό το οποίο ε, συνέταξε ο κ. Ντεπρέ για το θέμα μας. Αλλά να σας πω κάποια σημεία που με βρίσκουν ελαφρώς αντίθετο με το κείμενο. Ναι, χρειάζεται ολοκληρωμένη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν το δικαίωμα να κρίνουν το πόσοι θα μετεκατασταθούν στην επικρατεία τους. Και αυτή η συμβολή των 10.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό, το ΑΜΙΦ, αφορά το αρχικό κόστο της μεταγκατάστασης. Τα κράτη-μέλη γνωρίζουν καλύτερα το πόσους μπορούν να προστατεύσουν, να εντάξουν στην κοινωνία τους που είναι το πιο σημαντικό. Άλλο, Κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά την συμμετοχή στο ενωσιακό πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνεται σε προεδρική βάση. Πρόκειται για εγχείρημα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να συμφωνείτε. Επίση, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων κατάσταση ναι, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου ε, εγγύηση, κάποιο είδου υποστήριξη, αλλά δεν προβλέπεται. Οι εθνικέ ποσοστώσει ε, προσφύγων δεν καλύπτονται. Επίση, νομίζω ότι η εθνική, η συγγνώμη, η για του ε, πρόσφυγε έχει μακρά εμπειρία και θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, να την αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο σε σχέση με το ενωσιακό πλαίσιο. Οπότε, αυτά είναι τα πιο σημαντικά που ήθελα να σας τονίσω και θα συνεργαστούμε. Ο κύριος Κολυμέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ζερά Τεπρέ για την πολύ καλή του δουλειά. Στην έκθεση αυτή βλέπω μια κάποια συνέπεια σε σχέση με άλλες εκθέσεις ε, ε, που εξεργαζόμαστε. Παραδείγματο χάρη, διαδικασία σε ό,τι αφορά επικός των χωρών ή απάτριδων Έχουμε αναφέρει εκεί κάποια ποσά, 6.000 ευρώ ή και 10.000 ευρώ για τη χώρα που υποδέχεται έναν μετανάστη. Υπάρχει όμως και μια πρόταση της Κομισιόν όπου εκεί καταβάλλεται ένα επίδομα αλληλεγγύης 250.000 ευρώ. διακόπτει ο κύριος Δεπρέ. Θέλω να επαναλάβω αυτά που είπα στην αρχή της παρουσίασής μου. Εμείς δεν μιλάμε εδώ για το σχέδιο της ε, κατανομής των προσφύγων που θα αναθεωρήσει το σύστημα του Βουβλίνου. Οπότε δεν υπάρχει θέμα 250.000 και κυρώσεων, γιατί στην κατανομή των μεταναστών που έχουν των προσφύγων που έχουν φτάσει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούμε με ένα μηχανιστικό τρόπο να τους μοιράσουμε, σύμφωνα με ένα σύστημα που έχει προτείνει η Κομισιόν. Δεν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο εδώ. Εμείς μιλάμε εδώ για την μετεγκατάσταση που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λέει πως κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέτει έναν αριθμό ατόμων, 100.000 για παράδειγμα, που θα τους πάρει από τα στρατόπεδα που βρίσκονται γύρω από τις περιοχές σειράξεων για να τους επιτρέψει να έρθουν στα κράτη-μέλη. Και ο μηχανισμός και ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι αυτός, αλλά δεν υπάρχει υποχρέωση από, την, από τα κράτη-μέλη να δεχτούν συγκεκριμένον αριθμό. Αυτά αποφασίζουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν κυρώσεις και 250.000 ευρώ κτλ. Αν δεν δεχτούν τα άτομα αυτά, γιατί δεν είναι υποχρεωτική αυτή η ποσόστοση. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα μηχανισμό που λέει θέλουμε ένα στόχο ανθρώπων για μετεγκατάσταση και όποιο θέλει μπορεί να συμμετέχει. Τα 10.000 ευρώ θα σας πω τι είναι. Είναι το ποσό που στα πλαίσια τη εκτέλεσης αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος θα δίνουμε στα άτομα τα οποία θα μετεγκατασταθούν σε κάθε κράτο μέλο. Παράλληλα με αυτά μπορούν τα κράτη-μέλη μονομερώς να πάρουν την απόφαση για την μετεγκατάσταση και άλλων ανθρώπων εκτό του προγράμματο. Μπορούν. Μπορούν. Είναι δικό του θέμα εθνική κυριαρχία, αλλά δεν βλέπω γιατί πρέπει αυτό να πληρωθεί από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η πρότασή μου είναι να πούμε λοιπόν ότι παίρνουμε όσου εγγράφονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματο έτσι όπω προτάθηκε από αυτό το μηχανισμό. Για να μην υπάρχει παρανόηση. Εδώ δεν έχουμε καμία κύρωση. Καμία κύρωση. Γιατί δεν μιλάμε για την κατανομή. Και γι' αυτό σα διέκοψα και ζήτησα το λόγο. Συγχωρέστε με. Ευχαριστώ πολύ κύριε Συνάδε για τη συμπληρωματική αυτή παρατήρηση και επεξήγηση. Όχι, δεν θέλω να πάω στο υπόβαθρο. Πράγματι υπάρχει διαφορά, άλλη μια διαδικασία, άλλη άλλη. Α, όμως τα ποσά είναι διαφορετικά. Στη μία περίπτωση μιλάμε για 10.000 ευρώ, στην άλλη Και αυτό δεν το λέει η Κομισιόν ότι είναι κύρωση, ότι είναι ποινή αλλά ας, ως εισφορά. Και είναι τεράστια διαφορά. Τη μία έχουμε 10.000 ευρώ, την έχουμε 250.000 ευρώ. Φυσικά, ε, είναι σαφές. Όταν λέμε ότι πάμε σε ένα τρίτο κράτος και παίρνουμε απευθείας από τον καταβλισμό κάποιους πρόσφυγες. Συμφωνώ και ε, απόλυτα μάλιστα με τον κύριο Σάρβαμα ότι αυτό πρέπει να είναι θελοντικό. Η βάση πρέπει να είναι θελούσια και μπορούμε να δούμε για τα ποσά. Το θέμα είναι αυτά τα 250.000, μην τα ξεχάσουμε αυτά. Γιατί στην άλλη πρόταση περιλαμβάνεται αυτό το ποσό. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουν, ε, είναι αυθαίρετα ή όχι αυτά τα ποσά. Δεν πρέπει να είναι και τόσο αυθαίρετα. Από στρατηγικής πλευράς, πλευράς τακτικής, εγώ νομίζω ότι στην Επιτροπή Προπολογισμών θα πρέπει να μας απασχολήσει ακριβώς το ερώτημα. Ποιος είναι ο στόχος μας, τι θέλουμε να πετύχουμε. τέλο είναι σαφές ότι υπάρχουν διάφορα βήματα για τα οποία συζητούμε και που πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση και είναι όλα θετικά και ωραία. Η Ένωση πρέπει όμως επιτέλους να έχει μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. Δεν το έχουμε ακόμα αυτό. Γιατί δεν έχουν οριστεί ακόμη κάποιες πολύ σημαντικές παράμετροι και δεν φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη ε, είναι και τόσο πρόθυμα σε επίπεδο Συμβουλίου να συνεργαστούν και να προχωρήσουν. Πάντως πρέπει να ε, γίνουν κάποια βήματα, εμείς θα τα στηρίξουμε, θα ψηφίσουμε υπέρ, αλλά συνολική λύση δεν υπάρχει ακόμη. Δεν θα ήταν λοιπόν πιο συνεπές. Εντάξει, δεν είμαστε καθήλυνα αρμόδια επιτροπή βέβαια, όμως εμείς είμαστε η Επιτροπή που διαθέτει τα κονδύλια, εγκρίνει τη χωρίς των κονδύλιων, Μήπως να πούμε stop και ότι ναι θα δώσουμε τα κονδύλια όταν υπάρχει μια συνολική προσέγγιση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε. Αν αυτό είναι μέρος της δικής μας αρμοδιότητας. δεν θα πρέπει αντί να παρασυρθούμε από αυτή τη διαδικασία να ζητήσουμε με μετεπιτάσεως μία συνολική λύση. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητέ. Κύριε Ντεπρέλιο Πρόεδρο, αυτά τα 250.000, ξαναπείτε μα τελικά τι είναι, είναι κύρωση ή δεν είναι κύρωση. Είναι πρόστιμο. Ο κύριο Ντεπρέ. Δεν είναι το αντικείμενο της πρώτης φεστούμε, το ξέλεω και το ξαναλέω. Είναι το σχέδιο κατανομής για την τροποποίηση του συστήματος του Δουβλίνου, που λέει ότι το κράτος πρώτης εισόδου είναι αρμόδιο για την ε, επεξεργασία της αίτησης ναι. ασύλου. Και εκεί προβλέπεται ένα σχέδιο ε, κατανομής σχεδόν μηχανικό, το οποίο δεν θέλω να σχολιάσω μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπεται στο διατακτικό. Άλλοι το λένε πρόστιμο και άλλοι το λένε εναλλακτική εγώ προτιμώ αυτή την ε, δεύτερη διατύπωση. Γιατί αυτοί που δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το μηχανισμό το παρουσιάζουν ως κύρωση, ως πρόστιμο. Για να τα πω πιο γενικά λέει η Κομισιόν ή θα συμμετέχετε στο πρόγραμμα κατανομής ή στη χρηματοοικονομική αλληλεγγύη. Κάθε φορά λοιπόν που δεν δέχεστε έναν υπόλοιπο υποψήφιο που θα έπρεπε να πάρετε συνάρτηση με αυτό το σχέδιο κατανομής του μηχανισμού αναθεώρησης του Δουβλίνου, θα ε, βάζετε στο ταμείο 205.000 ευρώ. Αυτό αφορά την αναθεώρηση του Δουβλίνου, αλλά δεν μιλάμε για αυτό. Δεν μιλάμε για εισφορά ε, κάποιου κράτους μέλους. Μιλάμε για τον προπολογισμό της Ένωσης. Δεν υπάρχει υποχρεωτικός περιορισμός και υποχρεωτική συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα Αυτά τα 205.000 ευρώ, λέει ο πρόεδρος, από δημοσιονομικής πλευράς. Τι είναι, ήδη διπόροι, Από δημοσιονομικής πλευράς τι συμβαίνει ακριβώς. Ο κ. Ντεπρέ, από τεχνικής πλευράς, κύριε πρόεδρε, πρέπει να στραφείτε στην Κομισιόν να ρωτήσετε πώς γίνεται από τεχνικής πλευράς. Εγώ δεν το γνωρίζω. Πού, πού μπαίνουν αυτά τα ποσά στις τσέπες των κρατών στον ευρωπαϊκό Προεπολισμό δεν ξέρω αν με απατέμνει μου, ας μου τα πει η Κομισιόν καλύτερα. Νομίζω ότι πηγαίνει στο κράτος ε, που θα δεχθεί τον πρόσφατο που δεν δέχτηκε το άλλο κράτος. Σε αυτού τα ταμεία θα πάει το ποσό αυτό. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία για αυτό το μηχανισμό. Υπάρχει κάποιο από την Κομισιόν που μπορεί να επιβεβαιώσει αυτό που είπα ή όχι. Πρόεδρος. Αυτό το πρόστιμο, την κύρωση, όπως θέλετε πείτε το, πώς την αντιμετωπίζει η Κομισιόν. Ο κ. δεν έχει αποφασιστεί, δεν υπάρχει απόφαση ακόμα. Αν υπάρξει απόφαση, λέει ο κ. Ε, Άρτουι, από δημοσιογραφική πλευρά αυτό πώ το απεξεργάζονται. Είναι κάτι διαφορετικό, το ξέρω. Τι προβλέπετε λοιπόν να μας πει η Κομισιόν. Αν μπορεί παρακαλώ να απαντήσει. Αν έχει να δώσει μια απάντηση βέβαια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντεπρέ για αυτή την εντυπωσιακή άμυνα υπέρ της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το θέμα το πιο συγκεκριμένο προτιμώ να κάνω μια μικρή έρευνα και να επανέλθω μαζί μια γραπτή ε, απόφαση, με μια γραπτή απάντηση ώστε να σας έχω δώσει ορθά στοιχεία. Ωραία λοιπόν. Στην επόμενη συνάντηση η δική σας απάντηση Νομίζω πως όλοι όσοι ζήτησαν να μιλήσουν το έχουν κάνει. Κύριε Ντεπρέ, συμπερασματικά, η διάκριση λοιπόν κύριε Πρόεδρε να είναι ξεκάθαρη για να μην έχουμε παρανοήσεις για το φάκελο που έχουμε μπροστά μας. Θεωρώ φυσιολογικό να συνεχίσουμε τη σημερινή πρακτική που είναι πως όταν τα κράτη-μέλη εθελοντικά αποφασίζουν να συμμετέχουν στο ε, θέμα της μετακατάστασης να παίρνουν αυτά τα 10.000 ευρώ. Αν θέλει να είναι παραπάνω, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Εν πάση αυτό είναι στην πρόταση. Και απαντώ στον κύριο Κέλμαντ για την έλλειψη ευρωπαϊκή πολιτική. Να σα πω λοιπόν πω αυτή η μετεγκατάσταση όπω έχουμε σε αυτή την πρόταση είναι μια νόμιμη οδό έτσι ώστε για τα άτομα που έχουν ανάγκη διεθνού προστασία να φτάσουν στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με ασφάλεια. Η επιλογή των ατόμων που θα μεταγκατασταθούν θα γίνεται με την ύπατη αρμοστία του ΑΕΕ. Οπότε δεν μιλάμε για κάποιες αυθαίρετε δράσεις από κάποιον δημόσιο υπάλληλο που θα πάει επί τόπου. Όχι. Είναι μια νόμιμη οδός και είναι ο για τον οποίο στηρίζω αυτή τη διάταξη πολύ γιατί ο στόχος θα έλεγα τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι και το λέμε όλοι να μην είναι θύματα του τράφικινγκ, να μην πνίγονται στη Μεσόγειο και να μπορούν να φτάσουν νόμιμα και με διεθνή προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα υπόλοιπα έχουμε ανάγκη από άλλες διατάξεις, γιατί αυτή τη στιγμή κάποιοι πραγματικά διακινδυνεύουν ε, να χαθούν για να φτάσουν στις χώρες μας. Και γι' αυτό, για εκείνους δηλαδή, εδώ θα έχουμε την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Αυτό θα εφαρμοστεί. Μάλιστα. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι, λέει ο κύριο Σαρβαμά, αλλά θέλω να εξηγήσω με ποιο τρόπο βλέπω εγώ αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα για την επαναγκατάσταση όλων αυτών που θεωρούμε πως χωρίζουν διεθνούς προστασία. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό, με κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να ελαφρύνουμε κάπως τις πιέσεις που αντιμετωπίζουμε με το μεταναστευτικό και αν έχουμε ένα εκατομμύριο άτομα τα οποία συμπλήν θεωρούν πως πρέπει να εγκαταλείψουν μια χώρα γιατί δεν μπορούν να ζήσουν εκεί, γιατί είναι σε πόλεμο τότε με το συντονισμό της ΥΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να πάμε και να τους πούμε, κοιτάξτε, εμείς μπορούμε να πάρουμε 20.000 με επίγοντα τρόπο και με ένα συντονισμό, συντονισμένο τρόπο και με μια διαδικασία που ακολουθεί κοινά πρότυπα και που θα συμφωνήσουμε εμείς και αυτό ακριβώς συζητάμε να προχωρήσουμε την κατάσταση αυτών των ατόμων. Και μετά θα πρέπει να συζητήσουμε αν είναι το Συμβούλιο που θα κληθεί να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα μοιραστούν στα κράτη-μέλη. Δηλαδή σε 7.000 εδώ, 5.000 εκεί, 348 άτομα εδώ ή αν θα, αποφασίσουν, θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Τα κράτη-μέλη είναι εθολοντική η συμμετοχή τους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του σχεδίου κατανομής για όσους έφτασαν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία ή στην Ελλάδα, για παράδειγμα, και φτάσανε με τους γνωστούς τρόπους, γιατί στο μηχανισμό αυτό της μετεγκατάστασης ορίζει στόχους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο αποφασίζουν σε ποιο βαθμό θα συμμετέχουν. Τα κράτη-μέλη λοιπόν μπορούν να πούν θέλουμε ένα πέμπτο, ένα έκτο των όσων υπάρχουν εδώ στο τραπέζι. Αυτό που θα έλεγα είναι πως αυτό δεν θα πρέπει να μπερδευτεί με το πραγματικά αμφιλεγόμενο πρόγραμμα που έχει 250.000 κύρωση, πρόστιμο δηλαδή, γιατί δεν έχουμε επανεγκατάσταση των ατόμων που φτάνουν στα σύνορά μας. Και αυτό δεν έχει αποφασιστεί και δεν έχει περάσει καν από τα δικά μας τραπέζια. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Κύριε Όλτριχ. Uh, Νομίζω ότι τα όσα κάνουμε εδώ ως Επιτροπή Προϋπολογισμού είναι να προσπαθούμε να λύσουμε τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο. Δεν μπορούμε εμείς να το μοιράσουμε σε κομματάκια. Και παρόλο που έχουμε πολλέ πολιτικέ διαφορέ με τον κύριο Κόλμερ Καταλαβαίνω ποια είναι η άποψή του, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια κατάτμιση. Έχουμε στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν, γιατί ολόκληρη μεταναστευτική πολιτική, η πολιτική ασύλου, η πολιτική θεωρήσεων, γιατί αυτοί που θέλουν να φύγουν από τη Μέση Ανατολή μπορούν να ζητήσουν θεώρηση. Που φεύγουν και ζητούν βοήθεια και εμείς βοηθάμε τα κράτη-μέλη εθελοντικά αλλά διαφορετικά έρχονται παράνομα, μετά έχουμε τα 250. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την κατάτμιση και να τα μοιράσουμε σε διαφορετικά κομμάτια. Έχουμε μια εξαιρετικά πολυσύνθετη μεταναστευτική πολιτική που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία. Γιατί αν πούμε εδώ 10.000, εκεί 250.000, εντάξει, ποιο θα είναι ολόκληρο το σύστημα. Θα ανοίξει το σύστημα θεωρήσεων για όσου θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Εάν θέλουν και είναι έτοιμοι να πληρώσουν, θέλουμε να έρθουμε θεωρήσεις ή θέλουμε να πάμε στο στρατόπεδο και να φύγουν από τα στρατόπεδα επειδή θα τα πάρουν τα κρατημέλη. Πολλά. Και δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια κάνει πολύ σαφή συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική στο, στο Κοινοβούλιο. Διαφορετικά θα τα δούμε αποσπασματικά και θα προσπαθούμε να πούμε να, αυτό είναι το σύστημά μας. Ο κύριος Κέλμελ, ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάλι πάρα πολύ σύντομα ε, συνοψίζοντας. Ε, δείχνει η συζήτηση ότι αστικά βλέπουμε όλοι μας ε, το ίδιο πρόβλημα. Ε, καταλαβαίνω όλα όσα είπε ο συνάδελφος Ντεπρέ. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Έχουμε μία περίπτωση, έχουμε την εθελούσια υποδοχή κάποιων προσφύγων απευθείας από το τρίτο κράτος υπάρχει αυτά τα 10.000 ευρώ και ταυτόχρονα υπάρχει μια συζήτηση για μια άλλη πρόταση της Κομισιόν. Μεταξύ άλλων λέει, όταν έχει φτάσει ήδη κάποιος μετανάστης στην Ευρώπη, και αν υπήρχε, δεν υπάρχει ακόμα, αλλά αν υπήρχε, αν υπάρξει μια ποσόστοση κατανομής, εάν ένα άτομο δεν το πάρει η χώρα που θα έπρεπε να το πάρει, θα πρέπει να πληρώνει 250.000 ευρώ. Ποιος, ποιο κράτος θα ήθελε εθελοντικά άμεσα να πάρει έναν α, πρόσφυγα από ένα τρίτο κράτος. Εάν θα πρέπει ε, να δεχθεί υποχρεωτικά με βάση το σύστημα αυτό ποσόστοση κάποια άλλα άτομα που είναι ήδη στο τη Ένωση, ε, Αν δεν το κάνει θα πληρώνει 250.000 ευρώ. Επομένω, ποιο θα το διαλέξει ε, να το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε μια συνολική θεώρηση, ένα συνολικό κόνσεπτ γιατί τελικά αυτά τα μεμονωμένα μέτρα έχουν αντιπαραγωγικό, είναι αντιπαραγωγικά, αν τα δούμε έτσι απομονωμένα. Διευκρίνηση. Κύριε 250.000. Για κάποια χώρα που, που τις, δώσανε χίλιους και δεν τους δέχεται, ε, θα πάρει 500. Ντεπρέ. Αυτή η διάταξη είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή και εμείς σύντομα θα πρέπει να αποφανθούμε γιατί επίσης είμαι ο συντάκτης νομότης επ' αυτού. Και άρα έχω να πω ότι δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία για τα 250.000 ούτε από το Συμβούλιο ούτε από μας. Και να λέμε συνέχεια ότι δεν υπάρχει βούληση για μια συνεκτική πολιτική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ε, βλακία. Πρόκειται για εκατομμύρια το οποίο τρέχονται στα στρατόπεδα. Και επιβαρύνουν πάρα πολύ κάποιε χώρες όπως την Ιορδανία. Ε, Αυτή η πολιτική της ε, επανεγκατάσταση είναι το πώ θα πάνε σε κάποιε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τι αναλάβουν αυτέ οι χώρε και αυτό ο κόσμο να έχει κάποια δυνατότητα εξέλιξης στις χώρες που θα φιλοξενηθεί. Είναι η πραγματική κατάσταση. Και η μεταρρύθμιση του Δουβλίνου σε αυτό αφορά. Αυτή που ξέρετε με ποιες συνθήκες περνούν την Μεσόγειο ή τα Βαλκάνια όσο ακόμα μπορούν και έρχονται σε επικράτεια της Ένωσης όταν φτάνουν μέσα σε μια χώρα ή στα σύνορα και ζητούν άσυλο θα πρέπει Κανεί να διεκπαιρεώσει την αίτηση του άσυλου. Και τι λέει η συνήθιση ε, ε, ότι θα πρέπει να βρει εκεί πέρα ε, άσυλο, ε, δεν το λέει αυτό. Λέει ότι θα πρέπει η εξέταση της αίτησης να γίνει στα σύνορα. Μην τα ανακατεύουμε όλα. Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην πολιτική μας, αλλά θα πρέπει όμως να μην ξεχνούμε την πραγματικότητα όπως είναι, αλλά και τις διαδικασίες. Η συνθήκη πότε είναι του 51. Στην και της Γενέβης. Το 51 νομίζω λέει ο Πρόεδρος. Έγινε για να επιτρέψει αυτούς που θέλουν να φύγουν από τις κομμουνιστικές χώρες να έρθουν στην Δύση. Πρόεδρος. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο το πρόβλημα σήμερα. Άρα θα πρέπει να έχουμε μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση. Γιατί όταν λέμε για 10.000 ευρώ, ωραία. Αλλά ποιος είναι ο στόχος από πλευράς δημισιονομικής; Γιατί θα πρέπει να δούμε αύριο τι θα γίνει, τι θα λένε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Θα λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινή διαχείριση, ε, θα εκχωρήσει κάποιος ε, εθνική κυριαρχία. Ε, πώς θα αποφανθεί κάποιος για το βάσιμο της αίτησης ασύλου. Πολλές φορές παίρνει δύο χρόνια, παίρνει τρία χρόνια και μετά από αυτά τα τρία χρόνια εάν αποφασιστεί να μην του χορηγηθεί άσυλο του μετανάστη μα τότε μπορεί καν να μην τον θέλει η χώρα προέλευσης. αλλά είναι παράλογη κατάσταση. Προτίθενται επομένω ε, τα κράτη-μέλη να έχουν μια κοινή διαδικασία, μια προσταθμένες και ταχύτερες διαδικασίες, γιατί δεν είναι καν το θέμα τα 10.000 ευρώ απλώς. Νομίζω ότι ε, εμείς ως Επιτροπή Προϋπολογισμών να πούμε το, όλα αυτά ωραία, αλλά τι θα γίνει αύριο. Αν έχουμε ένα εκατομμύριο, ε, έχουμε τρία εκατομμύρια στην Τουρκία και αν το ένα εκατομμύριο από αυτούς έρθει θα σημαίνει ότι πάμε για ποσό 10 δις. Αυτό τι πάει να πει για τον προπολογισμό της Ένωσης να έχουμε σημειακά στοχευμένα μέτρα και αύριο να βρεθούμε σε δημισιονομικό αδιέξοδο γιατί το ε, Συμβούλιο δεν θέλει να συμπληρώσει, να κάνει το top-up, οπότε βρίσκεται σε μια θέση αδυναμίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να, πώς φουσκώνει ο λαϊκισμός. Σαρβαμά. Μα, ακριβώς αυτό λέμε, γιατί λέμε για λίγους, λίγους πρόσφυγες που δεχόμαστε. Ε, είναι το πιο σωστό να είχαμε μια συνολική, συνεκτική, πολιτική. Τι να σας πω, δεν θα πρέπει να λέω τέτοια πράγματα, αλλά πότε να γίνει κάτι τέτοιο, πότε θα θελήσουν τα κρατημέλη να πούνε «Οκ, okay, όλοι να ε, μοιραστούμε το βάρος εξίσου». Δεν είναι έτσι τώρα. τέλο πάντων για να διασκεδάζουμε τις αμφιβολίε, του, φόβου του Πρόεδρου. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να έχουν την αρμοδιότητα. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε με προσοχή να υπολογίζουν. Τι δεσμευτικές συμφωνίες συνάπτουν όσον αφορά την αναδοχή προσώπων από τρίτες χώρες και κατόπιν να λαμβάνουν τα 10.000 άτομα. Δεν νομίζω να φτάσουμε σε 100.000 για αυτή τη διαδικασία. Ε, τα είπε πάρα πολύ καλά ο κύριος Ντεπρέ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα, το resettlement, την επανεγκατάσταση και σίγουρα ε, θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τη συνολική πρόκληση. Ένα άλλο που θέλω να αναφέρω. Έχουμε την ε, συνθήκη 78, ε, μάλλον τα άρθρα 78-80 τη συνθήκη της Λισαβόνας και πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Ε, προσπαθήσαμε να υιοθετηθούν κάποιοι κανόνες, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το πρωτογενές δίκαιο ακόμη επαρκώς σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες επανεισδοχής της Ένωσης με τρίτες χώρες, ε, αν υπάρχουν ε, ιδιαίτερες καταστάσεις, ιδιαίτερες συνθήκες, ε, μπορούμε να αποφασίσουμε έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης. Και στο άρθρο 80 επίσης γίνεται λόγος για αλληλεγγύη και την δίκαιη ισομερία κατανομή των βαρών. Επομένως, μας δίνει το πρωτογενές δίκαιο όλες τις δυνατότητες αν δεν έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να έχουμε ένα πλήρε πακέτο μέτρων που θα αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα. Ωραία λοιπόν. Για να πάμε προς, ε, την, προς το τέλος της συζήτησης, γνωμοδότηση για μία πρόταση. Δεν είμαι ούτε ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε του, του Συμβουλίου. Εγώ απλώς προσπάθησα να το κάνω, να σας πω πάνω σε τι εργαζόμαστε ταυτόχρονα. Όσο δεν υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική μεταναστευτική και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το προσπαθεί. Αλλά υπάρχει μια σχεδόν απόλυτη, ε, ε, αδυναμία του Συμβουλίου να φτάσει σε κάτι τέτοιο. Αν λοιπόν το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχτεί τις προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να δείχνουμε ότι έχουμε συνοχή, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και θα μπορούσε να γίνει εδώ. Λοιπόν, δεν μπορεί να βρεθεί μια διατύπωση η οποία θα απευθύνει μια έκκληση στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πούν πιο συγκεκριμένα πως το μέτρο αυτό ε, ε, εντάσσεται σε ένα πιο ολοκληρωμένο όραμα και ότι εμείς θέλουμε να δούμε να μας δοθούν κάποια στοιχεία που θα μας εξασφαλίσουν πως οι δημοσιονομικές επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό δεν θα είναι τόσο βαριές. Εκτός μικροφώνου. Η Επιτροπή ΛΥΠΕ θα πρέπει να ε, σχολιάσει το πώς επηρεάζεται από τις προτώσεις αυτός ο προπολογισμό στην έκθεσή της. Προτείνω λοιπόν να μην κάνουμε τροπολογία, αλλά να πούμε ότι για το οικονομικό βάρος και την ανάληψη ευθύνης ε, να κάνουμε τη σχετική δήλωση. Θα πρέπει να πούμε πως είναι ο προπολογισμό του 18. Εκεί λοιπόν να το κάνουμε. Ναι, εμείς στην Επιτροπή Προπολογισμού δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα τέτοιο μεμονωμένο μέτρο χωρίς να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες για, την Ευρω... για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Γιατί θα μπορούσαμε με τον τρόπο αυτό να έχουμε πολλά έτσι μερικά προσπασματικά μέτρα, συμπαθητικά με, αλλά εμείς εξασφαλίζουμε πως υπάρχει συνοχή προϋπολογισμού και πως υπάρχει αυτή η δυνατότητα χρηματοδότησης των όσων έχουν αποφασιστεί. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι για να το κάνουμε έτσι, γιατί εγώ πραγματικά έχω έξω από τα ρούχα μου για το Συμβούλιο που δέχεται μόνο τα πιο βραχυπρόθεσμα μέτρα. Και κάθε φορά περιμένουμε να περάσουν κάποιες εκλογές. Αυτό δεν μπορεί να διονυστεί. μπορούμε κατά καιρού να εκφράζουμε ε, μια επανάσταση ε, ε, κατά αυτής της έλλειψης συνοχής γιατί δίνει μια πραγματικά θλιβερή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή ακριβώ η εικόνα είναι που τρέφει τον λαϊκισμό και την ανάγκη να κλείσουμε τα σύνορά μας και τα εδάφη μας. Λοιπόν, θα δω αν προτίσω εγώ κάποια τροπολογία. Δεν υπάρχει τροπολογία μάλιστα. Αντί να έχω τη δική μου γνωμοδότηση λοιπόν, μπορούμε να υποβάλουμε ένα ε, κείμενο. Μία αντίδραση. Μία αντίδραση πρέπει να εκφράσουμε. Γιατί εδώ διαφορετικά είμαστε στο αποσπασματικό. Δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Κύριε Φερνάντες. Τα γαλλικά μου δεν είναι καλύτερα από αυτά του Ζεράρντεπρε και δεν θα καταφέρω να τα εξηγήσω καλύτερα. Πολλά τα... Πολλά τα κομπλιμέντα που σας έχουμε κάνει, αγαπητοί συνάδελφοι. Όχι, αλλά το να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για την μετεγκατάσταση, εδώ είναι κάτι το πολύ διαφορετικό από την κατανομή. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις τροπολογίες. Συμφωνούμε λοιπόν με αυτή την πολιτική. Και θα μπορούσαμε να πούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι προφανώς πω δεν υπάρχουν πολλέ δημοσ... Ε, γιατί τα κράτη-μέλη εθελοντικά δεν αναλαμβάνουν αυτές τις ευθύνε. Αλλά υπάρχουν τέλο πάντων κάποιες δυνατότητε και ίσως για να κάνουμε κάτι πιο σφαιρικό, Και για το 2018 τον προπολογισμό το έχουμε ήδη κάνει και να πούμε θέλουμε κάτι πιο σφαιρικό, πιο, να δείχνει μεγαλύτερη συνοχή και να τα ε, θα επιτύσσουμε αυτά τις προσπάθειες που κάνουμε για τον προπολογισμό του 18 και όχι σε μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας που στο κάτω-κάτω είναι πάρα πολύ κλαδική. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Ζεράρ Ντεπρέ. Δεν συμβαίνει αυτό πάντα, αλλά σήμερα συμφωνώ απολύτω μαζί του. Μάλιστα. 11 η ώρα έφτασε. Ευτυχώς συμφωνήσαμε εγκαίρως, γιατί έχουμε την ώρα των ψηφοφοριών τώρα. Δεν έχουμε και πολλά να ψηφίσουμε. Αν εξελιχθούν τα πράγματα όπως τα φαντάζομαι, διότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό συμβάν, πολύ σημαντική εκδήλωση στην Ολομέλεια και επειδή κοστίζει ακριβά μια θέση στην Ολομέλεια, νομίζω ότι γύρω στις 11 και 10 θα πρέπει να είμαστε εκεί και όχι 11.30 για όποιον θέλουν να παρευρεθούν. Σε ευχαριστώ, Ζεράρια, για, τις, ε, για τη διαφωτιστικές σου επεξηγήσεις. Νομίζω ότι όλοι είχατε τη δυνατότητα να εκφραστείτε. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, θα απασχολήσει γενικότερα την Ευρώπη και στο πολιτικό επίπεδο. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού και Γενικός Εισηγητής για τον Προπολογισμό, ο κύριος Γέννης Γκάιρ, έχει το λόγο Μπορούμε να ψηφίσουμε, δεν έχω να πω κάτι. Έχω μόνο μία, γραμματεία, ε, μία ρόσπα γραμματεία για να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχουν ε, κάποια ασφάλματα σε ό,τι αφορά την τελευταία απόφαση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσωπής στην παγκοσμιοποίηση που έχουμε ε, επιτρέψει και κάποιες μεταφορές ε, πιστώσεων, αλλά αυτή τη συγκεκριμένη φορά δεν έχουμε να ψηφίσουμε για κάποια μεταφορά πιστώσεων. Τι υπάρχει να μας πει η γραμματεία. Δεν έχουμε να ψηφίσουμε λοιπόν, λέει ο πρόεδρος σήμερα κάτι. Τη Δευτέρα λοιπόν, αυτά που έχουμε εδώ. Sur la, la, justement, la mondialisation, ça fera l'objet. Για την παγκοσμιοποίηση ακριβώς πράγματι έχουμε να ψηφίσουμε, αλλά τη Δευτέρα. Και νομίζω απαντώ έτσι στο ερώτημα που έθεσε στη γραμματεία ο κύριος Γκάιερ. Υπάρχουν κάποιες αιτήσει μεταφορά σε άλλα τμήματα. Ο κύριος ε, Τάντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Όπω είδατε έκανα κάποια λάθη. Οπότε πρέπει να κάνουμε τώρα διορθώσεις με μεταφορές όλων πρώτα πρώτα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε εδώ αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πάρουμε κάποια χρήματα από τις ε, αμοιβέ και να τα πάμε σε κάποια νομικά εξόδα και αποζημίωση. Μιλούμε για 160.000 ευρώ, λέει ο κύριος Τάραντ, διότι κάποιοι Ευρωπαίοι κέρδισαν την δίκη των που είχαν προσφύγει. Αυτό είναι η πρώτη διόρθωση. Αυτή την μεταφορά πίστοσης προτείνω να την εγκρίνω. Ο πρόεδρος, αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, θεωρώ ότι εγκρίνεται την πρόταση, δεν βλέπω κάποιον να γεννήσει. Κύριε Γκρέσλε, συμπαθάτε με, αλλά δεν, δεν άκουγα για πιο πιο κονδύλι λέτε. Α, λέτε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ωραία, γιατί θέλω κάτι να πω. την πρώτη για την δεύτερη μεταφορά πόρων. Ήδη έχει ε, προηγηθεί κάποια την τελευταία φορά. Και να τα πω στα γερμανικά. Νομίζω ότι έχουμε αυτό το ποσό ε, το οποίο πρέπει να επιδικαστεί ε, σε βάρος του δικαστήριου που άρχισε να αποφανθεί, να βγάλει απόφαση. Νομίζω ότι δεν είναι καλό ούτε για το δικαστήριο, ούτε για την Ένωση γενικά να περιμένουν οι πολίτες τόσο πολύ ε, για την εκδίκαση κάποιας ε, υπόθεσης. Και πραγματικά τα πράγματα δεν βελτιώνονται. Νομίζω ότι θα πρέπει και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να καλέσει ε, τον γραμματέα του δικαστηρίου για να δούμε. Έχουμε άλλες παραλήψεις και καθυστερήσεις γιατί τον Φεβρουάριο είχαμε δύο αποφάσεις, ε, τρία δεν ξέρω πόσες ε, περιμένουμε ακόμη. Κέντριον κατά επιτροπής ήταν η μία οι δύο αυτές εταιρείε Πλάστικος Ισπανιόλες και Αρμάντο Αλβάρισταν, η δεύτερη και Γκασκόνια. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Γιατί τα πληρώνει ο ε, πολίτης αυτές τις καθυστερήσεις. Μήπως ε, ο εκπρόσωπος του δικαστήριου που είναι εδώ μπορούσε να απαντήσει. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ να σας πω ότι Έχουμε έρθει ήδη δύο φορές εδώ για να ζητήσουμε κάποια μεταφορά που είναι για φέτος, αλλά είχαμε κάποιο πρόβλημα καθυστέρησης της διεκπαιρέωσης των υποθέσεων στο δικαστήριο. Το 16. Οπότε θα πρέπει κατόπιν της ενίσχυσης του προσωπικού να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα στο μέλλον. Πάντως, είχαμε κάποιες ε, προσφυγές, αγωγές τέλος πάντων που υπευλήθησαν. Είχαμε τρεις καταδίκες φέτος και πρόκειται για ακόμα μια προσφυγή και τον επόμενο μήνα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση. Οπότε υπάρχει αυτό το θέμα της ε, υπέρβασης, της υπερβολικής καθυστέρησης τέλος πάντων της εκδόσης απόφασης απλώς στο δικαστήριο. Βεβαίω και στο μέλλον θα έχουμε και άλλες υποθέσεις που θα υποβληθούν στην κρίση του δικαστηρίου, αλλά προς το παρόν έχουμε μία, μία μόνο φορά ε, για την οποία θα πρέπει να προσφύγουμε στην Επιτροπή σας και να ζητήσουμε αυτή τη μεταφορά κονδυλίων. Ο πρόεδρος, α, μα το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν έχετε τα κατάλληλα μέσα, πόρους. Ε, δεν υπολογίσατε καλά το, ότι χρειάζεστε για να μπορέσετε να αποφασίσετε μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια. Θα πρέπει επ' αυτού να είμαστε σαφείς. Κύριε Γκρέσλα. Ναι, πράγματι. Το έχουμε ξαναπεί με το δικαστήριο. Θέλουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα της κατάστασης που δεν την έχουμε ακόμη, δεν έχουμε υπάρχει στοιχεία. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ολοκληρώνει εγκαίρως το έργο του. Θα πρέπει να οργανωθούν διαφορετικά Όλοι είμαστε υποποίηση και σε ό,τι αφορά το χρόνο μας και σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, το ε, προσωπικό. Το καταλαβαίνω. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να δούμε κατά πόσο είναι για ένα συγκεκριμένο τμήμα του δικαστηρίου, ε, ήταν το πρόβλημα η ανεπάρκεια δικαστών, κάπου αλλού ήταν το πρόβλημα και έχουμε πολλές άλλες υποθέσεις που θα καταδείξουν το ίδιο πρόβλημα ή όχι. Αυτό, αυτά όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ο κ. συνεχίζει. Συμφωνώ. Το πρόβλημα έχει όπως το διατύπωσε η κυρία Γκρέσλε. Και επί τη των στοιχείων που έχω, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι οι πόροι που λείπουν στο δικαστήριο οικονομική. Ε, πάντως το πρόβλημα είναι στην οργάνωση των εργασιών του. Βέβαια, τα κράτη-μέλη δεν τα πήγαν τόσο καλά στον διορισμό των νέων δικαστών όσον αφορά τις οικονομίες ε, που θέλαν να έχουν με το να μην, ε, να μην διορίσουν τους νέους δικαστές. Οπότε πρέπει να διορθωθούν τα λάθη τα λάθη τα οποία θα οδηγούν στη διώση των λαθών των κρατών στην εφαρμογή του δικαίου. Άρα, το θέμα δεν είναι το αν θα γίνει μεταφορά των πόρων από το ένα κονδύλι στο άλλο, αλλά το θέμα είναι ποιο θα πληρώσει του Γερμανού και Ισπανού ε, εμπορευόμενου επιχειρηματίε. Πάντω, συνάδελφοι, έτσι κι αλλιώ ε, σα ζητώ σήμερα να εγκρίνουμε αυτή την μεταφορά πόρων. Υπάρχει όμω και άλλο ένα θέμα που και του προπολογισμού και έχει δημοσιονομικέ επιπτώσει. Όταν το δικαστήριο λαμβάνει μια απόφαση με πρόστιμο προ μια επιχείρηση, τι γίνεται, εσπαράτεται αυτό από τον προπολογισμό έτσι ώστε να αποδοθεί στα κράτη-μέλη, στο εκείνο το κομμάτι του προπολογισμού. Όταν το δικαστήριο δεν καταφέρει να τελεσυδικήσει μέσα σε, μια, σε ένα εύλογο διάστημα, τότε ο προπολογισμό εισπράττει όχι τα κρατημέλη. Θα πρέπει λοιπόν το αποτέλεσμα των προστήμων που αποδίδονται στα κράτη-μέλη να δούμε τι γίνεται, γιατί αν ε, επιβάλλουμε κάποια κήρυξη στο δικαστήριο, το πρόστιμο αυτό αφαιρείται από τα ποσά τα οποία έχουν καταβάλει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όχι ο προπολογισμό. Μήπως θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μια τέτοιου είδους αρχή. Για τώρα, για φέτος ή για το επόμενο. <laughs> Όχι, για τα δύο. Γιατί το έχουμε συζητήσει, δεν είναι δίκαιο. Όταν πέφτει ένα πρόστιμο, το τσεπώνει το κράτος μέλος. Αν το δικαστήριο δεν αποφαίνεται έγκαιρα και υπάρχει κάποιο πρόστιμο, αυτό θα πρέπει να αφαιρείται από τα ποσά που έχει εισπάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, μια απλή υπόδειξη κάνω. Ο κύριος Γκάι. Άκουσα πολύ προσεκτικά και τελικά δεν ξέρω αν με αυτά που προτείνετε θέλουμε να αλλάξουμε ουσιαστικά ε, τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Όχι απόψε βέβαια. Ε, με την κυρία Γκρέσλε το έχουμε ξαναπροσπαθήσει. Τα κράτη-μέλη παίρνουν ε, στο τέλος του χρόνου ή θέλουν να πάρουν στο τέλος του χρόνου αυτά τα ποσά ε, και αυτά προβλέπει και η νομική βάση. Το θέμα είναι τι γίνεται με τη χρήση αυτών των ε, προστήμων και αυτών των ποσών. Όπως στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε αυτή την αμέλεια του δικαστηρίου. Είναι πολύ ειρωνικό που καταδικ... αυτό ουσιαστικά βέβαια το δικαστήριο, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι τι γίνεται ε, με αυτά τα χρήματα. Μπορώ να πάω στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο τιμωρείται ε, το δικαστήριο που παρέλειψε ή πάντων αμέλησε να αποφασίσει εγκαίρως. Αλλά αν εν λειτουργεί ένα όργανο όπως θα θέλαμε, ε, θα πρέπει να βγαίνουν κάποια χρήματα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα πρέπει να το δούμε. Σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, ποινές, αυτά τα πρόστιμα. Να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και όχι να τα βάζουμε στα ταμεία των κρατών μελών στο τέλος του χρόνου. Θα πρέπει να κλείσουμε την συνάντηση τώρα το συντομότερο, οπότε ο εισηγητής μας είπε να το ψηφίσουμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις. Εσείς είστε ε, ακόμα κατά. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε για την πίστοση αυτή ηλεκτρονικά νομίζω. Βλέπω όμως πως δεν έχω τη δική μου κάρτα μαζί, δεν είναι και σοβαρό. Ίσως η ανατάσεως της χειρός. Κύριε Ντεπρέ, ούτε εσείς έχετε κάρτα. Ποιος είναι υπέρ ε, αυτής της ε, μεταφοράς. Κατά. Ωραία, υπερψηφίστηκε. Δεύτερη μεταφορά που προτείνεται για την Επιτροπή Περιφερειών. Η πίστοση αυτή η Επιτροπή Περιφερειών. Προσπαθεί να εξορθολογεί όλο και περισσότερο το οργανόγραμμά της. Εδώ ζητείται μεταφορά πίστοσης για τη δημιουργία τροποποίηση κάποιων θέσεων, δεν ξέρω, νομίζω τα έχετε μπροστά σας, να μην σας τα διαβάσω ξανά. Το καλό νέο είναι ότι οι προτινόμενες αλλαγές δεν αλλάζουν το συνολικό αριθμό των θέσεων και υπάρχει και εξοικονόμηση της τάξης των 465 ευρώ και 70 λεπτών. Άρα νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη μεταφορά. Δεν χρειάζεται νομίζω να ψηφίσουμε, δεν νομίζω ότι πάει κάποια ένσταση. Επομένω έχουμε εγκρίνει τη συγκεκριμένη πρόταση για τροποποίηση κάποιων θέσεων. Θα διακόψουμε τώρα και στις 3 το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε, λέει ο πρόεδρος. Στις 3 λέει ο πρόεδρος. Α, με συγχωρείτε, διορθώνει ο πρόεδρος στις 2. Στις 2 το μεσημέρι. Η λέξη της συνεδρίασης.